Ladies and gentlemen. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο χρόνος τρέχει. Θα επαναλάβουμε την σύνοδο της ε, ΕΟΚΕ. Παρακαλώ καθίστε λοιπόν για να ξεκινήσουμε. Κυρίσω την έναρξη τη δεύτερη ημέρα ε, της συνόδου της ΕΟΚΕ και ως πρώτο σημείο με μεγάλη χαρά θα αφήσω το λόγο στη Μιλένα Αγγέλοβα που είναι αντιπρός, αντιπρόεδρος και πρόεδρος της ΚΑΦ της Ομάδας Προϋπολογισμού για να σας παρουσιάσει το σχέδιο προβλέψεων για τον προϋπολογισμό του 2020 που ομόφωνα το Προεδρείο ενέκρινε την Τρίτη το απόγευμα. Παρακαλώ Μιλένα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να τονίσω, όπως πολύ σωστά επισήμανε και ο Πρόεδρός μας, ότι η πρώην ομάδα του προπολογισμού έχει μετονομαστεί σε Επιτροπή για Οικονομικά και Δημοσιονομικά Θέματα, ΚΑΦ, και ε, έχει αυξηθεί κατά τρία μέλη, έναν ομάδα, και ελπίζω με τη νέα σύνθεση ε, που προβλέπουν ε, οι εσωτερικοί κανόνες, ο εσωτερικός κανονισμός, να εργαστεί η ΚΑΦ πιο αποτελεσματικά, ε, και να αξιοποιήσει το έπακρο του σπόρους μας. Θα ήθελα εν συντομία να σας παρουσιάσω την πρόβλεψη ε, δαπανών του προϋπολογισμού για το 2020 που ε, εγκρίθηκε από το Προεδρείο την Τρίτη και θα διαβιβαστεί στις 27 Μαρτίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σημείο αφετηρίας είναι οι προσπάθειες, οι μόνιμες προσπάθειες σε να, να προσαρμόσει τις προβλέψεις στις προσδοκίες όλων των ενδιαφερομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετά την κρίση κάνουν ε, μόνιμες εκκλήσεις για μέτρα λιτότητας και πολύ συνετή συμπεριφορά, κάτι που επηρεάζει αρνηστικά τον προπολογισμό μας. Από το 2015 διαπιστώνουμε ότι έχουμε μείωση σε πραγματικούς όρους 1,35% παρά το γεγονός ότι τα χρόνια αυτά ε, αν αυξήθηκε κατά 7,3% ο προπολογισμό μας, ε, ονομαστικά τουλάχιστον. Ταυτόχρονα, ο αριθμό του προσωπικού από 713 περάσαμε στου 668. Είχαμε μείωση του προσωπικού, 5% δηλαδή συνολικά μείωση του προσωπικού της ΕΟ και όπως είχα συμφωνήσει τα θεσμικά όργανα το 2013 και είχαμε μεταφορά 36 θέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει τη Συμφωνία συνεργασία. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μεγάλες πιέσεις στο έργο της ΕΟ και χάρη όμως στις ε, άγνες προσπάθειες της γραμματείας ε, του Γενικού Γραμματέα και όλων των συναδέλφων και μελών της ΕΟ και καταφέρουμε παρόλα αυτά να ανταπεξέλθουμε στο έργο μας. Κάθε χρόνο λαμβάνουμε επιστολή με τι βασικέ κατευθυντήρε γραμμέ Ευρωπαϊκή Επιτροπής, την επιστολή Έτιγκερ όπω είναι γνωστή, γιατί ο Επίτροπο Έτιγκερ είναι αρμόδιο, που δημιουργούν, δημιουργεί μάλλον το πλαίσιο για τι προ για τον επόμενο προπολογισμό. Για τον προπολογισμό του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω και στο παρελθόν, παρότρινε όλα τα θεσμικά όργανα να εφαρμόσουν ε, ένα ονομαστικό πάγωμα των προβλέψεών τους για όλες τις δαπάνε που δεν αφορούν μισθούς. Και ταυτόχρονα, η τη μαριθμική αναπροσαρμογή για του μισθού που ε, γίνεται θα γίνει τον Ιούλιο του 2019 και 2020 είναι 3,1% και 2,5% αντίστοιχα. Ο πληθωρισμός του από το Δεκέμβριο του 2018 μέχρι το 2020 αναμένεται σε 1,6% αυτός είναι ο υπολογισμός. Και όλοι όλα αυτά τα στοιχεία είναι η βάση των υπολογισμών μας και των προβλέψεών μας. Και οι συνάδελφοι της υπομάδας που κατέρτισαν τον προπολογισμό του 2020 και ο εισηγητής ο κ. Μεντόσα, στον οποίο είμαι ε, ιδιαίτερα ευγνώμων, καθώς και ο συναδέλφος Ρέμπερ και Ιμπάσκου, ε, κατάφεραν να αξιοποιήσουν στο έπακρο του σπόρους ε, δεδομένων των περιορισμών που αντιμετωπίζουμε και της συρρήκνωση του προϋπολογισμού. Οπότε τα έχουμε φροντίσει όλα, μπορώ να σας διαβεβαιώσω με ιδιαίτερη χαρά και έχουμε αύξηση κατά 4,22% του προϋπολογισμού μας ή 5,8 εκατομμύρια συνολικά και οι προβλέψεις μας για το 2020 είναι περίπου 144 εκατομμύρια, κάτι που υπολείπεται ε, τα 4,3% το κατόφλι δηλαδή που έχει τεθεί για την αύξηση του προϋπολογισμού όλων των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Εν συντομία λοιπόν αυτές είναι οι προβλέψεις του προϋπολογισμού μας για το 2020 και ελπίζω ότι θα εγκριθούν χωρίς περαιτέρω περικοπές. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ. Πάντως οι προβλέψεις μας είναι αρκετά συνετές και στερητικές και θα μας επιτρέψουν παρόλα αυτά να επιτελέσουμε το πολιτικό μας έργο. Σας ευχαριστώ. Thank you so much. Ευχαριστώ. Ε, δεν έχουμε τον έλεγχο της υποδομής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δυστυχώς, γιατί μερικές φορές έχουμε πόλεμο των μικροφώνων εδώ πέρα δεν ξέρουμε πώς να τα ενεργοποιήσουμε, να τα απενεργοποιήσουμε. Ευχαριστώ Μιλένα για την παρουσίαση. Δεν προβλέπεται συζήτηση, ήταν απλή παρουσίαση των προβλέψεων του προπολογισμού. Περνάμε κατευθείαν ε, στην εκνομοδότηση 612 του Σόκ. εκπαίδευση για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφύγουμε τις αναντιστοιχίες. Ε, η Μιλένα ε, Αγγέλα είναι η συγγήτρια, παρακαλώ έχετε το λόγο. Θα προσπαθήσω να σα κρατήσω ξυπνητού σήμερα το πρωί, κάτι που θα είναι εύκολο. Θα σα παρουσιάσω εν συντομία την έκθεση πρωτοβουλία για το τι αλλαγέ χρειάζονται για να προσαρμόσουμε τα εκπαιδευτικά μα στήματα και τα στήματα κατάρτισή μα στι προκλήσει τη αγορά εργασία και στι αλλαγέ των οικονομικών μοντέλων. Είμαι ευγνώμων στους συναδέλφου τη Ομάδα μελέτη που με υποστήριξαν και με βοήθησαν πολύ και λάβαμε υπόψη τις συζητήσεις που έγιναν στις τρεις τελευταίες προεδρίες γιατί η συγκεκριμένη γνωμοδότηση άρχισε να εκπονείται στα τέλη της Βουλγαρικής Προεδρίας, συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας και ολοκληρώνεται κατά τη Ρουμανική Προεδρία. Το μέλλον της εργασίας και της ψηφιοποίησης ήταν επίκαιρα θέματα και των τριών Προεδριών και ευχαριστώ επαναλαμβάνω και τις τρεις Προεδρίες που συνέβαλαν με τις προτάσεις τους και εμπλούτησαν τη γνωμοδότηση που πιστεύω ότι είναι ένα αξιόλογο έγγραφο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο μέλλον για να μας εξοπλίσει με καλύτερα εφόδια και ε, δεξιότητες. Διαπιστώνουμε ότι η αναντιστοιχεία δεξιοτήτων με τις ανάγκες αγοράς-εργασίας είναι γεγονός. Δεν πρόκειται να απαλλαγούμε από αυτές, θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη. Πάντως το επίπεδο ακόμη της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων είναι ανησυχητικό ακόμη. Κάτι που δημιουργεί στενοπού στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και εμποδίζει τους Ευρωπαίους πολίτες να αναπτύξουν το δημιουργικό τους δυναμικό και εμποδίζει και τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν στο έπακρο το δικό τους δυναμικό. Γι' αυτό χρειάζονται κάποια μέτρα. Οι αναντιστοιχεί αυτές των δεξιοτήτων επίσης ε, επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα στο σύνολο της κοινωνία, Εμποδίζουν ε, τους πολίτες να νιώσουν ε, ικανοποίηση με τη σταδιοδρομία τους και πολλές φορές συρρυκνώνουν τους μισθούς τους. Επίσης επηρεάζουν την επαγγελματική και οικονομική ανάπτυξη και περιορίζουν το ατομικό δυναμικό των εργαζομένων. Επίσης περιορίζουν την παραγωγικότητα κάποιοι υπολογισμοί έχουν δείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει 0,8 ευρώ ένα ώρα λόγω της αναδυστυχίας των δεξιότητων. Επίσης, ε, μειώνεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων με την επιβράδυνσή τους και την ε, αύξηση των δαπανών ε, σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση των ανθρώπινων πόρων ή τη διαφύλαξη των ανθρώπινων πόρων. Προτείνουμε λοιπόν κάποια απτά μέτρα για να ληφθούν απόψε από τα κράτη-μέλη και να προωθηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν, στον τομέα της επίσημης προειδοποίησης, α, της, συγγνώμη, της επίσημης κατάρτισης, αυτό πια δεν ισχύει. Ε, αλλάζει το μοντέλο και απαιτείται πια μια βασική εκπαίδευση που θα συνεχίζεται όμως διαβίου. Με μια διαβίου κατάρτιση και επιμόρφωση προκειμένου να εφοδιάζονται με τα κατάλληλα προσόντα και τις δεξιότητες οι εργαζόμενοι. Επίσης, το διαδίκτυο ε, απαιτεί λιγότερη ε, αποστήθηση, αλλά περισσότερη κριτική σκέψη, λύση προβλημάτων, ε, επεξεργασία πληροφορίας. Αυτές είναι τώρα οι ανάγκες και όχι τόσο η απομνημόνευση που ήταν στο παρελθόν γνώσεων. Εκτός από τις ήπιε δεξιότητε χρειάζονται περισσότερες δεξιότητε σε θετικές επιστήμες, μαθηματικά επι, ε, επιστημονικές ε, γνώσεις, τα STEM που λέμε, και επίσης θέλουμε και οι γυναίκες να προσεγγίσουν αυτές τις νέες ειδικότητε των θετικών επιστημών. Ε, των θετικών επιστημών. Θα πρέπει λοιπόν να αναπτυχθούν όλες αυτές οι δεξιότητες και να αξιοποιήσουμε τη θετική εμπειρία των πρωτοπόρων χωρών, της Γερμανίας και της Αυστρίας για παράδειγμα, που έχουν πολύ καλές επιδόσεις σε τέτοιες επιτυχίες. Επίσης, το πανεπιστημιακό πτυχίο δεν είναι πια κανένα χέγγιο επιτυχίας. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε καλύτερη ενημέρωση του κόσμου με σωστές πληροφορίες, ώστε να κάνουν τεκμηρωμένα και περιστατωμένα τις επιλογές τους και να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους. Σας ευχαριστώ. Thank you so much. So the list is closed. Μάλιστα, ολοκληρώνει το κατάλογο στον ομιλητό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σας συνάδελφοι. Θα ήθελα να συγχαρώ τη Μιλένα για την αρτιότατη γνωμοδότησή της που πραγματεύεται ένα τεράστιο πρόβλημα της μοντέρνας εποχής τι αναντιστοιχίε των δεξιοτήτων με τι απαιτήσει αγορά εργασία. Θα πρέπει λοιπόν να σκοπωθούν τα κράτη-μέλη και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά του συστήματα και τα συστήματα κατάρτιση στι νέε ανάγκε. Επίση, θα πρέπει να αποκρινόμαστε συνεχώ και να προσαρμοζόμαστε στι αλλαγέ. Οι εξελίξει είναι ραγδαίε στην τεχνολογία. Η κατάσταση μεταβάλλεται αλλεπάλληλα και θα πρέπει και εμεί ε, να είμαστε πιο ευέλικτοι για να προσαρμοστούμε καλύτερα αξιοποιώντα τι βέλτιστε πρακτικέ και τα καλά παραδείγματα. Πολύ καλή λοιπόν η γνωμοδότηση. Και είναι καλό να γίνονται εκτενείς συζητήσεις στην Ολομέλεια σε τόσο καλές γνωμοδοτήσεις. Στόχος της γνωμοδότησης που κατέθεσα με τον κύριο Τράντινα, τον Μπάβελ Τράντινα, ε, μιλούμε για την τυπική και άτυπη επιμόρφωση ε, και παραπέμψαμε σε μια προηγούμενη μας γνωμοδότηση. Αυτό είναι το περιεχόμενο της τεχνικής ουσιαστικά τροπολογίας που υποβάλαμε. Πάντως, στόχος μας είναι να γίνει εκτενή συζήτηση αυτής της γνωμοδότησης, γιατί είναι τόσο καλή που της αξίζει να προβληθεί όσο γίνεται. Ευχαριστώ η Τατιάνα Μπαμπραουσκένε για δύο λεπτά. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη Μιλένα γιατί είχα τη χαρά να είμαι πρόεδρος αυτής της ομάδας μελέτης και χαίρομαι που κατάφερε ε, να συμπεριλάβει με ισορροπημένο τρόπο όλε τις απόψεις τη γνωμοδότησή της. Μάλιστα ζήτησε και τρίτη συνεδρίαση εξέτασης γιατί λόγω απεργιών στι στις Βρυξέλλες δεν μπόρεσαν όλοι να εκφέρουν τις απόψεις τους και δεν κατάφεραν να έρθουν στη δεύτερη συνεδρίαση, γι' αυτό έγινε και τρίτη. Η Μιλένα λοιπόν κατάφερε όχι μόνο να καταρτήσει μια πολύ άρτια και ισορροπημένη γνωμοδότηση, αλλά έπιασε το πνεύμα αυτή τη δύσκολη εποχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε τόσε προκλήσει, τόσο ρηξικέλευθο μετασχηματισμό τη οικονομία μα εντόπισε την ανάγκη μεταρρύθμισης και των εκπαιδευτικών μας συστημάτων και της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και των <clears throat> προγραμμάτων κατάρτισης. Οι δεξιότητες θα είναι το κλειδί για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις τεράστιες προκλήσεις. λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, λόγω της αλλαγής των οικονομικών και επιχειρησιακών μοντέλων, λόγω της αλλαγής των μοντέλων απασχόλησης και εργασίας. Ευχαριστώ θερμά, Μιλένα, για τη γνωμοδότησή σου. Ελπίζω να την αξιοποιήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Ευχαριστώ. Thank you. And now, Pavel Ευχαριστώ, κύριο Στραντίνα, το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια για την εξαιρετική περιγραφή των προκλήσεων που συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση της. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι στα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης είναι αναγκαίο να μπορεί κανείς να έχει την ευελιξία και όσον αφορά την αναγνώριση και όσον αφορά τη μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο. Αναφερθήκατε στις ε, ήπιες δεξιότητες ή τις διατομεακές διεπιστημονικές δεξιότητες. Αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι η παράγραφος 3.3, η οποία αναφέρει ότι αν κανείς έχει πανεπιστημιακό πτυχίο, αυτό βεβαίως δεν μπορεί να σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να συνεχίσει την ε, διαβίου μάθησή του. Αντιθέτως, η διαδρομή αυτή επεκτείνεται και παρατείνεται κατά τη διάρκεια και της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός ανθρώπου. Και αυτό αναφέρεται επίσης και στην παράγραφο 1.8 και όπως ε, είπε και η συγγήτρια, εδώ ε, νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια να ξεκαθαριστούν κάπως τα πράγματα. Πέρσι ήταν η προθεσμία ε, έως την οποία τα κράτη-μέλη ήταν υποχρεωμένα να παρουσιάσουν τα εργαλεία τους για την αναγνώριση δεξιοτήτων και προσόντων που έχουν αποκτηθεί εκτός του επίσημου τυπικού ε, εκπαιδευτικού συστήματος. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλομορφία μεταξύ των κρατών μελών. Είναι μια τεχνική τροπολογία, αυτή που έχω καταθέσει και θεωρώ ότι εμπλουτίζει την έκθεση στο σύνολο της. Ευχαριστώ πολύ, Μιλένα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, συνάδελφοι, για τα καλά σας λόγια και για την κατάθεση τροπολογιών που μας έδωσε τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτή την ε, έκθεση σήμερα το πρωί. Τις δέχομαι τις τροπολογίες γιατί ε, νομίζω ότι τονίζει και τον ρόλο των ε, εκπαιδευτικών ε, ιδρυμάτων Συγγνώμη, κατάλαβα, ε, λέει ο Πρόεδρος, ότι δέχεστε τις τροπολογίες. Υπάρχει κάποιος που αντιτίθεται στις ε, τροπολογίες αυτές. Όχι. Οπότε γίνονται αποδεκτές και περνάμε κατευθείαν στην, ε, στην ψηφοφορία για την ΣΟΚ 576 της κυρίας Μιλόβα. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is ψηφοφορίας. 134 ψηφίσαντες, μόλις δύο ε, αποχές, 130 υπέρ, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, και περνάμε στη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, Stop στον Εξτρεμισμό. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Ράιμερ και τον κύριο Λάιουπς από την Οργανωτική Επιτροπή αυτής της ε, Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας. Φτάνουν εδώ στο βήμα. Θα ξεκινήσω εγώ με μια μικρή εισαγωγή στο θέμα. Κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε, τον Απρίλιο, σε λίγες μέρες δηλαδή, θα εγκριθεί από τους δύο συνομοθέτες ο νέος κανονισμός για τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών. Αυτό το σημαντικό στοιχείο της συμμετοχικής δημοκρατίας. Κάτι που θα συμβάλλει στην διευκόλυνση της συλλογής υπογραφών για τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες. Είναι καλά τα νέα αυτά για την Ευρώπη και κυρίως για τους Ευρωπαίους πολίτες. Και χαίρομαι πάρα πολύ που οι δύο συνομοθέτες κατάφεραν να καταλήξουν σε συμβασμό ώστε να ε, τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία πριν από τις ευρωεκλογέ. Γιατί αυτό θα δώσει πλέον τη δυνατότητα στους πολίτες με ευκολότερο τρόπο να εκφράσουν τις γνώμεις τους, να υποβάλουν τα αιτήματά τους και να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως Επιτροπή είμαστε χαρούμενοι και πολύ περήφανοι για αυτή την εξέλιξη. Γιατί ως, όπως γνωρίζετε η ΕΟΚΕ έχει κάνει κάθε προσπάθεια ακόμη και πριν από την ε, υιοθέτηση της συνθήκης Λισαβόνας, για να προωθήσει αυτήν την ε, ε, δυνατότητα των πολιτών να συμμετέχουν άμεσα στην δημοκρατική διαδικασία και καλέσαμε πολλές φορές να υπάρξει η θέσπιση αυτού του εργαλείου, αυτού του μηχανισμού. Στην τελευταία μας γνωμοδότηση για την πρόταση της Κομισιόν, η κυρία Κιγκαγιού είχε τονίσει την προσήλωση της ε, ΕΟΚΕ και την επιθυμία της να είναι ε, συστατικό στοιχείο αυτής της διαδικασίας. Ξέρετε ότι κάθε χρόνο ε, εμείς οργανώνουμε την ημέρα για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών όπου δίνονται πληροφορίες, γίνεται ένας απολογισμός για το τι έχει αποφέρει θετικά αποτελέσματα και τι όχι τόσο θετικά αποτελέσματα. Η φετινή ημέρα ε, για άλλη μια φορά θα έχει αυτόν τον ε, στόχο, αυτόν τον χαρακτήρα. Θα ε, προσέλθει μάλιστα στην εκδήλωση αυτή και ο κύριος Τίμερμανς που θα παρουσιάσει τους νέους κανόνες στις φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε και τη δυνατότητα στα μέλη μας να συμμετάσχουν, να σε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Ράιμερ, Σιμπάστιαν Ράιμερ και τον κύριο Μίχαελ Λάουψερ, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν σήμερα την πέμπτη επιτυχή Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Στόπ στον εξτρεμισμό». Μια πρωτοβουλία που 12 μήνες μετά την έναρξή της έχει ε, έχει καταφέρει να συγκεντρώσει 1,6 εκατομμύρια υπογραφές. Αυτή τη στιγμή οι υπογραφές επαληθεύονται από τα κράτη-μέλη, αλλά πραγματικά ο αριθμός αυτός είναι εντυπωσιακό. Βασικός στόχος ε, αυτής της πρωτοβουλίας είναι, είναι προφανώς, προφανής και από, την, ε, από τον τίτλο της και θα έχουμε σήμερα την ευκαιρία να συζητήσουμε εν ώψη και των ευρωεκλογών αυτό το θέμα, εν ώψη των κινδύνων που εμφανίζονται μπροστά στι ευρωεκλογέ για την άνοδο του εξτρεμισμού. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σήμερα η ΕΟΚΕ για άλλη μια φορά είναι το πρώτο θεσμικό έργο, ε, όργανο που δίνει το λόγο σε πολίτες που έχουν ε, τεθεί επικεφαλής μιας τέτοιας ε, πρωτοβουλίας που θα εξεταστεί μόλις ολοκληρωθεί η επαλήθευση των υπογραφών. Θα δούμε τώρα ένα μικρό βιντεάκι στο οποίο θα μπορέσετε να δείτε τα βασικά επιτεύγματα και το βασικό θέμα αυτής της πρωτοβουλίας και στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στους πολίτες που έχουμε σήμερα μαζί μας και ήταν επικεφαλής αυτής της πρωτοβουλίας και στη συνέχεια θα γίνει και συζήτηση με τα μέλη. Παρακαλώ να δούμε το βίντεο.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 We need a million supporters. We need you. Support us and sign the initiative today. Dear Mr. President. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την πρόσκληση που μας απευθύνατε για να σας παρουσιάσουμε σήμερα εδώ την Πρωτοβουλία Πολιτών. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, συγχαίροντας την επιτυχία μας, θα πίστευε κανείς ότι έπρεπε να είχαμε φέρει σαμπάνιες, αλλά δυστυχώς βρισκόμαστε ακόμα στη διαδικασία επαλήθευσης των υπογραφών. Πράγματι, έχουμε συλλέξει πάνω από 1,6 εκατομμύρια υπογραφές πολύ περισσότερες δηλαδή από όσες χρειάζεται. Πρέπει όμως να επαληθευτούν και γι' αυτό είμαστε ακόμα αρκετά προσεκτικοί ε, σχετικά με το νομικό αποτέλεσμα της ε, πρωτοβουλίας μας. Προτού ο συντάκτης αυτής της πρότασης οδηγίας ε, της πρωτοβουλίας ε, Stop στον εξτρεμισμό σας παρουσιάσει μια μικρή σύνοψη πρότασης οδηγίας Θέλω να σας δώσω μια σύντομη επισκόπηση σχετικά με την πρωτοβουλία που αναλάβαμε και τι έχουμε επιτύχει. Η πρωτοβουλία Stop στον είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών η οποία αποσκοπεί στο να θέσει ένα τέρμα σε αυτήν την κόποση που εμφανίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αντιμετώπιση του εξτρεμισμού από την αριστερά, τη δεξιά και από θρησκευτικές ε, ομάδες. Θέλουμε λοιπόν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συζητήσουν από κοινού το πώς μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις εξτρεμιστικές, ε, αυτά τα εξτρεμιστικά φαινόμενα που συμβαίνουν εδώ στην Ευρώπη. Δεν χρειάζεται νομίζω να αναφερθώ και στα γεγονότα της Νέας Ζηλανδίας ε, ή της Ουτρέχτης ε, αυτή την εβδομάδα. Πραγματικά είναι επιτακτική ανάγκη να αναλάβουμε δράση. Και αυτό είναι και το βασικό περιεχόμενο της πρωτοβουλίας μας. Όπως είπα και νωρίτερα, ε, σκοπός μας είναι η καταπολέμηση του ακροαριστερού, του ακροδεξιού εξτρεμισμού, του εξτρεμισμού που έχει θρησκευτικά κίνητρα, της ρητορική μίσους ε, στον πραγματικό και στον ηλεκτρονικό κόσμο. Και αυτό αυτός είναι ο σκοπός ε, της πρώτας οδηγία μας. Θέλω να αναφέρω ότι το μίσος έχει αρχίσει και πραγματικά δημιουργεί ρογμές ε, στις κοινωνίες μας. Το κράτος δικαίου, δικαίου παίζει όλο και λιγότερο ρόλο στην θεσμική και πολιτική μας συζήτηση. Ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων χρειάζεται να υποστηριχθεί ε, περισσότερο, ιδίως από τις ε, κοινωνίες της Ευρώπης. Η επιρροή από χώρες και ομάδες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται. Γίνονται τρομοκρατικές επιθέσεις. Και εδώ βλέπετε κάποια στατιστικά στοιχεία σχετικά με τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν από την 11η Σεπτεμβρίου. Τα δεδομένα αυτά, τα στοιχεία αυτά είναι από το 2017. Βλέπετε λοιπόν ότι οι Ισλαμιστικές τρομοκρατικές επιθέσεις ε, δυστυχώς βρίσκονται πάνω-πάνω στον κατάλογο αυτό. Στη συνέχεια έχουμε τον ακροδεξιό εξτρεμισμό, αλλά και άλλα είδη. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα υπερκομματικό ευρωπαϊκό υπόδειγμα ε, το οποίο θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός αυτής. Επίσης, θα σας τα πει και ο Σεμπάστιαν, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ξένη χρηματοδότηση εξτρεμιστικών δομών. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ξένα ε, κέντρα να χρηματοδοτούν ε, φορείς εδώ στην Ευρώπη. Από την μουσουλμανική αδελφότητα έως το 2017 είχαν μεταφερθεί 120 εκατομμύρια ε, ευρώ, σε ευρωπαϊκούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Χρηματοδοτήθηκαν τζαμιά όπου διδασκόταν ο εξτρεμισμός και ο φονταμενταλισμός και θέλουμε να ζητήσουμε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αυτή, ε, και να τους επισημάνουμε το γεγονός ότι όταν ο εξτρεμισμός συνοδεύεται από χρήματα είναι πιο επικίνδυνος από τον φτωχό εξτρεμισμό. Οπότε πρέπει πραγματικά να αντιμετωπίσουμε αυτήν την χρηματοδότηση. Η ξένη χρηματοδότηση πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και ζητούμε να θεσπιστούν και κυρώσεις σε περίπτωση που ε, πραγματοποιούνται παράνομες ε, μεταφορές χρημάτων, χρηματοδοτήσεις. Επίσης, να αναφέρω το γεγονός ότι ο ορισμός του εξτρεμισμού είναι δύσκολο να, να, να είναι ένας ορισμός στον οποίο θα συμφωνούν όλοι. Εμείς ε, ισχυριζόμαστε ότι εξτρεμισμός είναι όταν κάποιος ενεργεί με τρόπο που θέλει να καταργήσει τα θεμελιώδη δικαιώματα που ε, συμπεριλαμβάνονται στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτός που κάνει κάτι τέτοιο, που ενεργεί έτσι, πρέπει να θεωρείται εξτρεμισμός. Μηδενική ανοχή στον εξτρεμισμό, λοιπόν. Και αυτό είναι το βασικό σημείο της, πρωτοβουλία, της πρωτοβουλίας μας που θα σας περιγράψει και ο Σεμπάστιαν. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι παρούσα και να υπάρχει και στο μέλλον και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Για να γίνει αυτό, η Ευρωπαϊκή, ερώτηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει απαντήσεις εκεί όπου τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να το κάνουν. Εξτρεμισμός, τρομοκρατία, ακροδεξιός εξτρεμισμός, ρητορική μίσου Όλα αυτά είναι φαινόμενα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο. Μπορεί, μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο σε πολυεθνικό, ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πιστεύουμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα της μπορούν να αποκτήσουν και την εμπιστοσύνη των πολιτών αν προβεί σε τέτοιες ενέργειες. Το γεγονός ότι 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι υπέγραψαν την πρωτοβουλία μας αποδεικνύει ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση. Και αυτό είναι αυτό που ζητάμε κι εμείς. Πρωτού μπω σε κάποιες λεπτομέρειες, θέλω να σας παρουσιάσω τον Ζεμπάστιαν Ράιμερ, που είναι νομικός και είναι ο συντάκτης ε, ολόκληρης της πρωτοβουλίας πολιτών στο στον Σα Σας δίνω το λόγο. Um, Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία και την τιμή που μου δίνετε να σας κάνω αυτήν την εισήγηση. Ε, πράγματι είμαι νομικός, ε, έχω ξεκινήσει από το γραφείο της καγκελαρίας στην Αυστρία αφού σπούδασε βεβαίως ε, νομικά διότι υπήρχαν ευκαιρίες για τους νεότερους διοικητικούς υπάλληλους ε, μια διαδρομή που ξεκίνησε από το υπόγειο γραφείο της καγκελαρίας ε, όπου εδώ και πολλά χρόνια διεξάγονται αυτά τα προγράμματα κατάρτισης γνωρίζουμε από την αυστριακή ιστορία ότι στον ίδιο χώρο παλαιότερα πραγματοποιούνται ε, εκτελέσεις εχμαλώτων και νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα συνεργασίας με έναν θεσμό, έναν φορέα, την καγκελαρία δηλαδή, γιατί αντιλαμβάνεται κανείς καλύτερα τι είναι αυτό το οποίο προασπίζεται. δίνουμε αγώνα στην Ευρώπη, έχει χυθεί αίμα, ώστε να προστατεύσουμε αυτά τα δικαιώματα που έχουμε εγγράψει στο χάρτη. Έχουν καταβληθεί λοιπόν πραγματικές προσπάθειες, διαβάζοντας ε, τις εφημερίδες, τον τύπο, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αντιμετωπίζουμε ένα κρίσιμο πρόβλημα, έχουμε βίαιο εξτρεμισμό. Όλοι είδαμε τις ε, φρικαλές εικόνες από το Christchurch, από τη Νέα Ζηλανδία, ε, οι οποίες χρησιμοποιούνται προπαγανδιστικά ώστε να δημιουργηθούν νέοι εξτρεμιστές για να εκδικηθούν. Δηλαδή ο ακροδεξιός ε, ακτιβισμός, ο φασισμός και ο ακραίος Ισλαμισμός είναι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος, λέει ο μιλητής. Εμείς δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηροί. Θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση σύμφωνα με την παράδοσή μας, σύμφωνα με τον πολιτισμό μας. Οι μόνες απαντήσεις που μπορούμε να δώσουμε είναι μέσω του φιλελευθερισμού, του κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λόγος για τον οποίο συνέταξα αυτό το κείμενο εγώ δεν ήμουν ποτέ πολιτικοποιημένο στο παρελθόν, αλλά αυτά τα φαινόμενα με όθησαν στο να αναλάβω την πρωτοβουλία αυτή που δεν ήταν καθόλου εύκολο έργο και υψηλού κινδύνου. Ε, το 80% των ανθρώπων που συναντήθηκα το τελευταίο 1,5 χρόνο ήταν υπό αστυνομική προστασία, που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Δηλαδή εμεί δεν συναντηθήκαμε με τους εξτρεμιστέ, συναντηθήκαμε με αυτούς που είχαν υψώσει το ανάστημά τους κατά των εξτρεμιστών, όπως φιλελεύθεροι μουσουλμάνοι. Αυτό ήταν ο λόγο τον οποίο συνέταξε αυτήν την οδηγία για να δοθεί μια λύση. Καταρχάς, ώστε να έχουμε έναν σαφή ορισμό του τι είναι εξτρεμισμός. Το κοινό, οι πολίτες, οι νομοθέτες, οι αστυνομικές αρχές δεν μπορούν να δράσουν παρά μόνο αν γνωρίζουμε και συμφωνούμε για το τι είναι εξτρεμισμός. Μέχρι στιγμής έχουμε μια στατιστική προσέγγιση η οποία δεν μας καλύπτει. Στην περίπτωση που έχουμε μια δεξιά στροφή στην κοινή γνώμη, γιατί παραδοσιακά ασχολούμασταν με ακροαριστερές οργανώσεις, λέει ο μιλητής. Δίνουμε λοιπόν έναν ορισμό πλέον του εξτρεμισμού με βάση το περιεχόμενο. Εάν πλήττει κανεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, ορίζεται ω εξτρεμιστή με βάση την οδηγία αυτή. Αυτό που φοβούνται όλοι οι εξτρεμιστέ είναι η διαφάνεια. Εμεί εισήγαμε διατάξεις επαρκούς νομικής και δικονομικής προστασίας για τους πολίτες και υπάρχει και ένας κατάλογος που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο που δίνει την ευκαιρία στους εργοδότες ε, στα σχολεία <clears throat> μεταξύ άλλων να απομακρύνει τους εξτρεμιστές, να προστατευτεί από αυτούς. Ε, μέσω ενός μείγματος ε, θετικής όθησης και αποτροπής. Αν δεν θέλετε δηλαδή να βρίσκεστε σε, έναν κατάλογο, σε μια μαύρη λίστα, τότε δεν πρέπει να συμμετέχετε σε φαινόμενα, σε δραστηριότητες εξτρεμιστικές. Αυτή είναι η αποτρεπτική πλευρά. Και εδώ έχουμε εκπαιδευτικά ιδρύματα, κοινωνικές οργανώσεις, ε, δημόσιες αρχές, όλους εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες, όλοι αυτοί που εργάζονται προς την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να λαμβάνουν μια πιστοποίηση. Το γνωρίζουμε ως διαδικασία μέσω των ε, βιολογικών ή οργανικών ε, τροφίμων. Σας ενδιαφέρει λοιπόν πού πηγαίνουν τα παιδιά σας στο σχολείο. Φαντάζομαι ότι όλοι οι γονείς θα ήταν πιο ανακουφισμένοι εάν είχαν ένα πιστοποιητικό που να λέει ότι δεν σημαίνει τίποτα περίεργο ή κακό στο σχολείο αυτό. Αυτά είναι θετικές προτροπές. Να έρθω λίγο στον ορισμό του εξτρεμισμού όλα ξεκινούν συνήθως με τα μηνύματα μίσους που είναι πολύ επικίνδυνα φαινόμενα διότι μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης φτάνουν σε μεγάλες ομάδες του κοινού. Βεβαίως και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για θετικό σκοπό τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά μπορούν δυστυχώς να χρησιμοποιηθούν και έτσι και είναι πολύ ισχυρό εργαλείο. Ο εξτρεμισμός λοιπόν πλήττει τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουμε συμπεριλάβει 27 συγκεκριμένες περιπτώσεις προκειμένου να διαφωλύνουμε την εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Έχουμε τα μηνύματα μίσους, έχουμε τις εκστρατείες κατά της εκπαίδευσης, κατά της παιδείας που είναι και αυτές οι φοβερά επικίνδυνες. Δεν ξέρω πόσες θέσεις απασχόλησης έχουμε σήμερα, θα έχουμε σε 5 σε 10 χρόνια, αλλά φανταστείτε τι θα γίνει αν η ανεργία ανέλθει. Αυτό δεν θα είναι καθόλου καλό για την πολιτική σταθερότητα, λέει ο μιλητής. Έχουμε περιπτώσεις ε, διακρίσεων στο δικαστικό σύστημα όπως στα ποινικά συστήματα της Σαρία. Έχουμε υποστήριξη προς τα εξτρεμιστές, συνεργασία και βεβαίως χρηματοδότηση. Τέλος βεβαίως, σας είπα για τη θετική προτροπή που είναι η πιστοποίηση, έχουμε τον ουδέτερο ορισμό του εξτρεμισμού και έχουμε την αποτροπή που είναι η watch list, αυτός ο κατάλογος, και είναι και οι χρηματικές κυρώσεις. Η οδηγία αυτή δεν ορίζει ποινές κράτησης γνωρίζετε την ιστορία του Αμπου Ghraib. Ο καλύτερος τρόπος να δημιουργήσετε αποφασισμένους εξτρεμιστές είναι να τους βάλετε στη φυλακή μαζί με άλλους τέτοιους. Και τότε μαθαίνει ο ένας τον άλλο και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Το πρόβλημα είναι εάν οι εξτρεμιστές είναι καλά χρηματοδοτημένοι και προέρχονται αυτές οι οικονομικές ενισχύσεις από διάφορους πόρους, το πράγμα καθίσταται ακόμα πιο, πιο περίπλοκο. Εγώ έχω μια εμπειρία στην νομοθεσία προστασία δομένων και είχαμε πραγματικά αρνητικότατε εξελίξεις τα τελευταία χρόνια σε αυτό το επίπεδο με τον ε, κανονισμό προστασίας των δεδομένων ιδιαίτερα ε, σχετικά με την ισότητα των φύλων αλλά γιατί να εστιαστούμε σε ένα θεμελιώδες δικαίωμα αν διαβάσει κανεί το άρθρο 54 που είναι από τα πιο σημαντικά της χάρτα, λέγει ότι δεν μπορεί να πλήττεται το ένα θεμελιώδες δικαίωμα ε, μέσω τη επιχειρηματολογία υπέρ άλλου. Πρέπει όλα τα δικαιώματα αυτά να προστατεύονται ταυτόχρονα την ίδια στιγμή και με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει λοιπόν να δούμε την ε, αποδυνάμωση των άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και αυτό το κάναμε. Έχουμε αποζημίωση και απλουστευμένη αποζημίωση που απορρέει από την νομοθεσία για τις διακρίσεις. Έχουμε πολλά καινοτόμα στοιχεία στις σελίδες της οδηγίας και θα, είχα, θα μπορούσα να σας την αναλύσω σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε κάποια άλλη ευκαιρία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Thank you both for Ευχαριστούμε και τους δύο για την παρουσίαση, λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε τον Πρόεδρο της ομάδας 2, Όλιβερ Ρότκε, για, δύο, για τέσσερα λεπτά από την Αυστρία και αυτός. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα. Αγαπητέ κύριε Ράιμα και Λάουψ, εκ μέρους της ομάδος εργαζομένων να σας καλωσορίσω και εγώ στην ΕΟΚΕ στον οίκο της κοινωνίας των πολιτών με τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Νέα Ζηλανδία είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή, πιστεύω, να σκεφτούμε πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον εξτρεμισμό, τα μηνύματα μίσους, τη βία που απορρέει από τέτοιες ε, αρνητικές ιδέες. μιλούμε για την ε, για την πόλωση της κοινωνίας μας και αυτό είναι ένα φαινόμενο, αυτές οι περιχαρακωμένες θέσεις είναι ένα φαινόμενο που πλήττει όλες τις χώρες. Και πρέπει να καταπολεμήσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Με την άνοδο επίσης ε, ακραίων πολιτικών κομμάτων και θέσεων. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και αυτή ευάλωτη σε αυτό. Εμείς ως ομάδα εργαζομένων είχαμε συμφωνήσει με την UNESCO ότι δεν είναι επαρκή να αντιμετωπίζει κανείς τον εξτρεμισμό απλώς. Πρέπει να τον αποτρέπει. Αυτό ξεκινάει από τα σχολεία. Δίδοντας μέσα στους μαθητές να αυξάνουν την αντοχή τους έναντι των μηνυμάτων αυτών, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που καταλήγουν στην απομόνωση και στον εξτρεμισμό. Πρέπει να βελτιώσουμε τη δυνατότητα όλων των πολιτών να συμμετέχουν ισότιμα, δίνοντάς τους και την ελπίδα ε, καλά αμοιβόμενων ε, θέσεων εργασίας, δηλαδή απόλυτη ένταξη στην κοινωνία. Πέρυσι, στο τέλος του έτους, η Επιτροπή υιοθέτησε μία γνωμοδότηση για την αποτροπή του τρομοκρατικού περιεχομένου online. Σχετικά δηλαδή με τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούν οι τρομοκρατικές οργανώσεις και πώς μπορεί η δίωξή τους να είναι πιο αποτελεσματική. Τι πρέπει δηλαδή να κάνει το κράτη-μέλη προκειμένου να υπερασπιστούν το κράτος δικαίου και να έχουν μηδενική αντοχή στα μηνύματα μίσους και τα φαινόμενα βίας. Online αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά και συχνά έχουν ε, απτές συνέπειες στην πραγματική ζωή. Έχουμε καταχρήσεις στο διαδίκτυο για να διαδοθούν, να διαχυθούν μηνύματα μίσους παντού στον πλανήτη. Πρέπει να εξακολουθούμε να υπερασπιζόμαστε την ελευθερία έκφρασης και πρόσβαση σε επαρκή ενημέρωση για όλους τους πολίτες. Γιατί τα μέτρα κατά του εξτρεμισμού δεν πρέπει ποτέ ε, να καταλήγουν στην απαγόρευση της έκφρασης. Δεν πρέπει δηλαδή να πλήξουμε τις ίδιες τις αξίες και αρχές που υποτίθεται ότι υπερασπιζόμαστε, δηλαδή το κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη και την ελευθερία έκφρασης. Θα ήθελα λοιπόν και πάλι να σας ευχαριστήσω για την ε, εισήγηση, για την παρουσίαση και για τη συζήτηση αυτή. Ελπίζω ότι η πρωτοβουλία σας θα ε, συνεισφέρει γιατί μόνο μέσω του διαλόγου ε, θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε, Όλιβερ. Και τώρα ο Τσίλιαν Λόν από την Ιρλανδία για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την παρουσίαση. Θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ κάτι στη συζήτηση. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές για το ποια είναι τα αίτια του εξτρεμισμού και τη ανόδου του λαϊκισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Είχαμε μια α, κατάρρευση του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού μα συστήματο. Και η λύση για την κατάρρευση αυτή ήταν η ανασυγκρότηση του ίδιου συστήματος που μας οδήγησε στην καταστροφή και να το χρηματοδοτήσουμε με μια διαδικασία λιτότητας, με τη χρήση των πολιτικών λιτότητας, γιατί απλοί εργαζόμενοι και οι βιοπαλαιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλήρωσαν ένα άδικο τίμημα για να περισσώσουν ένα σύστημα που κατέρευσε και δεν τους είχε εξυπηρετήσει καν. Και έχουν περάσει 10 χρόνια από την έναρξη της κρίσης και το μήνυμα που λαμβάνουμε από τους ηθήνοντες ε, σε εξουσίες είναι ότι βρισκόμαστε σε φάση οικονομικής ανάκαμψης. Και ε, υπολογίζαμε το GDP, την, ε, το ΑΕΠ, δηλαδή την ανάπτυξη, την δανειοδότηση, με τρόπο που να, μας, να προσπαθεί να μας πείσει ότι επιτύχαμε και έχουμε οικονομική ανάκαμψη. Αυτό όμω που βιώνουν οι πολίτες είναι κάτι τελείως διαφορετικό, γιατί οι πολίτες βλέπουν άλλους δείκτες όπως τη φτώχεια, όπως τους αστέγους την μετανάστευση τα προβλήματα με τη διάβρωση του εδάφους, τις κλιματικές αλλαγές. Οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί δείκτες περιγράφουν μια πολύ διαφορετική εικόνα από τους ε, ε, οικονομικούς δείκτες που γίνονται π.χ. τίτλοι και βρίσκονται στο φως της δημοσιότητας. Η πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες ε, δεν ανταποκρίνεται στα λογίδρια και στους δείκτες που μας παρουσιάζουν οι, οι και οι κατέχοντες στην εξουσία, τα λόμπι, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, ε, ο οικονομικός κλάδος ε, αποκλίνουν από την πραγματικότητα των πολιτών. Κάτι που δημιουργεί πρόσφορο και γόνιμο έδαφος για τον εξτρεμισμό, τον λαϊκισμό, τα fake news, την παραπληροφόρηση, γιατί ε, έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους, γιατί άλλα βιώνουν και άλλα ακούνε ως πραγματικότητα οι πολίτες και αυτό τους αποσταθεροποιεί. Όλα αυτά δημιουργούν γόνιμα έδαφο λοιπόν για τον εξτρεμισμό γιατί μόνο στον εξτρεμισμό βρίσκουν ε, κάτι για να ταυτιστούν μερικές φορές οι Ευρωπαίοι πολίτες. Γι' αυτό θέλουμε το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσουν τα εφόδια που έχουν και τα εργαλεία που έχουν για να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα και κυρίως το θέμα των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης για να επανισορροπήσουμε και πάλι τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα με τις οικονομικές ανάγκες, λαμβάνοντα υπόψη τα δικαιώματα των πολιτών και τη φύση και να τα δούμε στο πλαίσιο της οικονομίας. Αν δεν γίνουμε ρεαλιστές ε, για την ανάγκη πραγματική συστημικής αλλαγής και αν δεν χρησιμοποιήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη ως μοντέλο για κάτι τέτοιο, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε τις βαθύτατες ε, αιτίε αυτών των φαινομένων. Ευχαριστώ, Τζίλιαν. Ο Γκονσάλο Ξαβιέ από την Πορτογαλία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω πορτογαλικά. Οπότε φορέστε τα ακουστικά σας. Σας ευχαριστώ για αυτά που μας είπατε και την πρωτοβουλία που αναλάβατε. Η πρωτοβουλία αυτή, κατά τη γνώμη μου, καλά, ε, ξεκινά. Είναι μια θετική πρωτοβουλία και έχει ένα θετικό μήνυμα. Και τα θετικά μηνύματα είναι, κατά τη γνώμη μου, ε, μια λύση για να πούμε stop στον εξτρεμισμό. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι πολλά από αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη, γιατί για την Ευρώπη μιλούμε σήμερα κυρίως εδώ, γίνονται ε, γιατί δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να, να σταματήσουμε τον το αυτομαστίγωμα και τον αυτοακροτηριασμό λόγω των λαθών του παρελθόντος. Παρελθοντολογούμε υπερβολικά και μαστιγωνόμαστε αντί να κοιτάμε προς το μέλλον με ένα θετικό μήνυμα. Αυτό είναι το σωστό. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει μία και μόνη συνταγή για να σταματήσουμε τον εξτρεμισμό και τον ριζοσπαστισμό. Υπάρχουν όμω τρόποι ζωή που βοηθάν τον πολίτη να αναγνωρίσει την αξία τη κατάσταση του και να ε, συμμετέχει στην κοινή ζωή, στη ζωή τη κοινότητα για να έχει πλήρη οικονομική, κοινωνική συγγνώμη, ένταξη. Γιατί αυτό χρειαζόμαστε, μια πλήρη κοινωνική ένταξη. Μόνο έτσι θα ξεριζώσουμε τον εξτρεμισμό. Είμαστε Ευρωπαίοι και διαβιούμε σε ένα χώρο που έχει το καλύτερο βιωτικό επίπεδο στον πλανήτη. Έχουμε ένα κοινωνικό σύστημα που έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Θα πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε την αξία αυτής της κατάστασης. Και ως ε, πρόσωποι των εργοδοτών αντιμετωπίζουμε και αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας στα θέματα της δημιουργίας και της ε, κατανομής του πλούτου. Σίγουρα η Ευρώπη δεν έχει ούτε μία εταιρεία στις 10 καλύτερες, στις 10 σημαντικότερες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου. Και στην Ευρώπη σίγουρα χάσαμε κάπως την ανταγωνιστικότητά μας. Αυτή όμως η ανταγωνιστικότητα δεν εγκατέλειψε την κοινωνική ευμάρεια, δεν εγκατέλειψε το βιωτικό επίπεδο, την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, την ανάπτυξη και ένα κοινωνικό μοντέλο που είναι το καλύτερο κοινωνικό μοντέλο του κόσμου αυτό που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάσαμε λίγο στην οικονομική μας ανταγωνιστικότητα ίσως, αλλά συνεχίζουμε παρόλα αυτά και παρά τις αντίξωες συνθήκες να ε, διαθέτουμε το καλύτερο κοινωνικό μοντέλο στον κόσμο. Ε, και αυτό περνάει από την εκπαίδευση στα σχολεία, από την ανάγκη να αναδεικνύουμε τις ευρωπαϊκές αξίες, την αξία της οικογένειας, που είναι πολύ σημαντική, την ε, ζωή της κοινότητας, τη δικαιοσύνη, την ειρήνη. Γιατί σήμερα ζούμε σε έναν κόσμο όπου η ελευθερία είναι μια αναπαλωτρίωτη αξία. Αλλά δυστυχώς δεν ζουν όλοι ελεύθερα. Εμείς στην Ευρώπη ζούμε ελεύθερα. Και μερικές φορές δεν εκτιμούμε την αξία αυτής της ελευθερίας. Γι' αυτό και είμαστε τέτοιο πόλο έλξη μεταναστών, χάρη στην ελευθερία που εξασφαλίζουμε. Αυτή η ελευθερία όμω θα πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλου. Και λέω σεβαστή και όχι να, μην επιβάλλεται. Ε, ελευθερία για αυτό που τρώμε, για την πίστη που πρεσβεύουμε, για το αυτοκίνητο που αγοράζουμε. Ε, και δεν θα πρέπει αυτή η αξία να χρησιμοποιηθεί για ιδιωτελείς σκοπούς. Και σίγουρα ε, το στόπ στον εξτρεμισμό περνάει από την ελευθερία των μειονοτήτων αλλά και από την ελευθερία των πλειονοτήτων, την ελευθερία για όλους. Γι' αυτό και χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία και χαιρετίζω και το θετικό της μήνυμα γιατί στην Ευρώπη και με την Ευρώπη θέλουμε να συνεχίσουμε να διαβιούμε και με το δικό της κοινωνικό μοντέλο. Σας ευχαριστώ. Obrigado. Η Τσίντι Αντελερίο από την Ιταλία για τρία λεπτά τώρα. Ευχαριστώ τον Σεμπάστιαν και τον Μίκαελ ε, για την παρουσίαση της ε, πρωτοβουλίας και αυτή την νομική προσέγγιση, αν θέλουμε να έχουμε έναν ορισμό του εξτρεμισμού. Βεβαίως η δουλειά τώρα ξεκινάει, δεν ολοκληρώνεται με αυτή την πρωτοβουλία, τη χρειαζόμαστε την πρωτοβουλία αυτή κατά του εξτρεμισμού που πλήττει τα θεμέλια του ευρωπαϊκού εγχειρήματο, αλλά χρειαζόμαστε άμεσα μηνύματα και οδηγίες για να καταπολεμούμε κάθε μορφή εξτρεπισμού, ιδιαίτερα στα πλαίσια αυτής της προεκλογικής εκστρατείας για τις ευρωπαϊκές εκλογές και προερχόμενη από μια χώρα όπου χρησιμοποιείται πολύ ο λαϊκισμός, ο εξτρεμισμός υποβοηθείται πολλές φορές από την ε, πολιτική σκοπιμότητα της στιγμής, όπως συμβαίνει στη χώρα μου σήμερα, με λαϊκιστικές επιθέσεις και πολιτικάντικα μηνύματα θα έλεγα, ε, ανθρώπων που φιλοδοξούν να εκπροσωπηθούν ε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και σημαίνει την καταπολέμηση και των μηνυμάτων ξενοφοβίας, ρατσισμού, νεοφασισμού, νεοεθνικισμού, δηλαδή τάσεων που βλέπουμε να διαχέονται ιδιαίτερα ε, ενεργητικά τον τελευταίο καιρό. Ε, τα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Μία έννοια είναι ο σεβασμός των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ένα άλλο θέμα είναι ο, ο σεβασμός και, τελεία. Δηλαδή να μην τοποθετούμαστε με τρόπο που πλήττει την διαφορετικότητα που είναι και αυτό θεμέλιο της δημοκρατίας. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο πνεύμα και να μην κλείνουμε τη ματιά μας και την ε, πολιτική μας τοποθέτηση πρέπει να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη αλληλεγγύης και συμπερίληψης με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, τους κοινωνικούς φορείς, δηλαδή ένα κίνημα για τη δημοκρατία που θα πρέπει να ξεκινάει από τους πολίτες, από την κοινωνία και όχι από την κορυφή και από την ηγεσία ώστε να ανακτήσουμε και αυτό το πνεύμα του διαλόγου που κάπως έχουμε απολέσει. Σήμερα να θυμίσω ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συζητούμε για μια πρόταση που αφορά την καθημερινή ζωή των πολιτών. Εχθές στην Ιταλία κοντά στο Μιλάνο έγινε μια απόπειρα κατά ενός σχολικού με 50 ε, παιδιά, μαθητές ο οποίος ε, διαμαρτυρόταν ένας εξτρεμιστής τα έκανε αυτά που διαμαρτυρόταν για τις ε, ανθρώπινες ζωές που χάνονται στη Μεσόγειο. Υπάρχει όμως και εξτρεμισμός ε, των λεγόμενων και όχι μόνο των παραξενών όπως έλεγε η Τσίνσια και τα ακούμε όλα αυτά τα λόγια, αυτούς τους λόγους, τους διαδρόμους του Κοινοβουλίου στη χώρα μας ε, ο υπουργό Εσωτερικών Σαλβίνη είναι ο ηγέτης αυτής της ορολογίας που χρησιμοποιείται ε, μηνύματα που μπορούν να οθήσουν στη βία υπάρχει εξτρεμισμός ε, και συμβολικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε φαινόμενα με επιθέσεις σε νεκροταφεία από νεοναζιστές και νεοφασιστές βλέπουμε ε, να προσπαθούν να δώσουν με διαφορετική ερμηνεία σχετικά με ιστορικά περάσματα επιθέσεις κατά των Εβραίων που είχαμε στη χώρα μας. Έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα σε ανατολικές χώρες, στην Πολωνία ιδιαίτερα και στην Ουγγαρία, όπου ε, πλήττεται η ανεξάρτητη δικαιοσύνη και ο ανεξάρτητος τύπος ε, αυτά είναι επικίνδυνες επιθέσεις η τροπή πάντοτε καταγγέλει και προσπαθεί να επιβάλλει κυρώσεις τα τραστ αλλά είναι πολύ πιο αφηρημένη και καθυστερή όταν πρόκειται για κυβερνήσεις κρατών μελών που πλήττουν την ελευθερία, τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ελευθερία των πολιτών κινείται πολύ γρήγορα όταν μιλούμε για οικονομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα, κινείται πολύ βραδέω όταν μιλούμε για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Ευχαριστώ, Αντώνιο Διακόπτη, ο Πρόεδρο. Ο Στεφάν Τουρτό τώρα από τη Γαλλία για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα του εξτρεμισμού είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, αλλά ταυτόχρονα και λεπτό. Οι κοινωνίες μας έχουν ξαναγίνει βίες κοινωνίες, κάτι που είχαμε ξεσυνηθίσει. Ε, η εφημερίδα Le Monde υπολογίζει ότι πέρυσι 3.000 άνθρωποι ήταν θύματα ισλαμιστικών ε, ε, ενεργειών στον κόσμο. Οπότε έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια κινήματα που θεωρούν ότι η βία είναι μια θεμητή έκφραση θεμητή έκφραση απόψεων. Αυτό ισχύει για, τον Ισλαμιστικό, για την Ισλαμιστική τρομοκρατία, για αυτά που συνέβησαν στο Παρίσι την, το προηγούμενο Σαββατοκυριακό. Θα πρέπει όμως να είμαστε σαφείς, γιατί ακούμε σε διάφορες ανταποκρίσεις και ρεπορτάζ για τα γεγονότα του Παρισιού ε, της περασμένης ε, εβδομάδας, ε, σε ένα κτίριο που φλέγεται μία γυναίκα με την κόρη της βρίσκεται στον όροφο ε, και λένε ότι θα κάψουμε τους πλουσίους από κάτω, ορίονται τα πλήθη. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση όπου έχει νομοποιηθεί ε, το μίσος και η βία από αυτούς που την ασκούν. Αυτός είναι ο εξτρεμισμός. Η νομοποίηση της βίας ως τρόπου δράσης. Γίνεται πια θεμητή η βία. Ε, είχα ζήτηση με τον δήμαρχο των Βεσσαλιών, ε, ο Μοχαμέτ Μεράντα ε, πυροβόλησε εξ παιδιά Εβραίων σε μια συναγωγή. Εξ επαφής σκότωσε παιδιά αυτός ο δράστης. Τι άνθρωπος είναι αυτός που διαπράττει μια τέτοια ενέργεια. Είναι άνθρωπος ή χάνει αυτή την ανθρωπιά πια. Επίσης, μερικές φορές Έχουμε ε, κάποιες ε, απόψεις που μπορεί να είναι ισχυρές. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει οι εκφράζοντες αυτή την άποψη να σέρνονται στα δικαστήρια. Είναι σημαντικό να έχουμε ελευθερία έκφραση. Τώρα, ό,τι αφορά τα πιστοποιητικά. στη Γαλλική Επανάσταση που είχαμε μια περίοδο ε, μεγάλης βίας, 17.000 άνθρωποι έπεσαν στη Λεμιτόμο, 3.000 γυναίκες, μιλώ για τις υπόλοιπες φαγές. Εκεί τότε είχαμε πιστοποιητικά ε, φρονήματος. Όσοι δεν είχαν τέτοια ε, πιστοποιητικά φρονημάτων έπεφτε στη λεμιτόμο. Προσοχή λοιπόν με τα πιστοποιητικά. Και εμείς έχουμε ένα μητρό που περιλαμβάνει τους ε, τρομοκράτες, Ισλαμιστές και άλλους. Είναι συσημασμένοι. Και μερικές φορές η δικαιοσύνη και η ασφάλεια βλέπουν αυτό το μητρό τόσο σημασμένο, αλλά από τη στιγμή που δεν έχουν περάσει στα έργα, δεν μπορούν να φυλακίσουν κάποιον επειδή μόνο είναι Ισλαμιστή, επειδή είναι φασιστή ή επειδή είναι αναρχικό. Οπότε υπάρχει μια έμπρακτη δυσκολία καταπολέμησης της, του εξτρεμισμού. Και η πρωτοβουλία σα με κάποια σύνδεση όμω θα μπορούσε να είναι μια αφετηρία ενδεχομένω. Ευχαριστώ, Στέφαν η τελευταία παρέμβαση από την κυρία Ζενεβιέφ Σαβίνη από τη Γαλλία επίσης. Καλημέρα σας. Θα μιλήσω στα γαλλικά. Είμαι μέλο τη ομάδα 3 για τη διαφορετικότητα στην Ευρώπη. Και με θάρρη να αναλάβω το λόγο στη συζήτηση, γιατί εγώ δεν κατάλαβα το νόημα αυτής τη πρωτοβουλία των πολιτών και δεν κατάλαβα τον όρο που χρησιμοποίησατε. Και έκανα κάποιε έρευνε. και ε, δεν διαφωτίστηκα γιατί μερικές ιστοσελίδες λειτουργούσαν καν. Αναφερθήκατε στον εξτρεμισμό αλλά και στην εσωτερική αγορά. Δεν κατάλαβα από αυτά που διάβασα στην έρευνα που έκανα για την πρωτοβουλία σας. Μετά τη συζήτηση άρχισα να ξεκαθαρίσω κάπως τα πράγματα, αλλά εξακολουθώ να διαβλέπω κάποιες απειλές σε αυτή την πρωτοβουλία. Κάποιες απειλές εις βάρος των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ακούσαμε σήμερα και χθε. <coughs> δηλαδή την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα του ανθρώπου, τη δημοκρατία, την ελευθερία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα, τη διάκριση των εξουσιών και το κράτο δικαίου. Κάποιε τέτοιε αξίε απειλούνται, όπω η ελευθερία έκφραση, το δικαίωμα να διαφωνεί κάποιο με τι κρατούσε οικονομικέ και πολιτικέ κατευθυντήριε γραμμέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το δικαίωμα να εκφράσει τη διαφωνία του. Η ιδέα ότι η λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι τέτοια με συνθήκε που έχουν αξία συντάγματο, ενώ υπάρχουν πολλοί άριθμοι πολίτε που καταδικάζουν αυτέ τι αξίε, ασκούν κριτική, ε, θέλουν να τι τροποποιήσουν, καταγγέλουν την πολιτική λιτότητα και τον αθέμητο ανταγωνισμό απέναντι σε χώρε που δεν έχουν του ίδιου κοινωνικού κανόνε, κάνουν dumping, δεν έχουν την ίδια φορολογία, δεν έχουν τι ίδιε αρχέ ίδιες ε, για τη χρήση φυτοφαρμάκων, για παράδειγμα, εντομοκτώνων, για να αναφέρω μερικά παραδείγματα. Καλώ κάναμε κάποιε διευκρινήσει, αλλά θα πρέπει να διευκρινίσουμε ακόμη περισσότερο την έννοια του εξτρεμισμού, να είμαστε πιο ακριβείς. Αν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε κάποια κινήματα ξενόφοβα, ρατσιστικά, εξτρεμιστικά, εντάξει. Αν θέλουμε όμω να εμποδίσουμε οποιοδήποτε κοινωνικό κίνημα, οποιαδήποτε κριτική, οποιαδήποτε ε, αφισβήτηση των κανόνων του παιχνιδιού, περιθωριοποιώντα και αποκλείοντα πολλού ευρωπαίου πολίτε, τότε έχω πολλού ενδιασμού για αυτή την πρωτοβουλία. Και αυτό που προέχει είναι να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, τη κοινωνική ανισότητα. Αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα του εξτρεμισμού. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Εν κατακλείδη, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά όλους ε, όσοι έλαβαν το λόγο για τη συμμετοχή τους. Να ευχαριστήσω θερμότατα τους οργανωτές αυτής της πρωτοβουλίας, γιατί περάσατε από τα λόγια στα έργα. Γνωρίζουμε ότι όταν προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τον εξτρεμισμό, ελοχεύει ο κίνδυνος δημιουργίας νέου εξτρεμισμού. Αλλά η πρωτοβουλία σας νομίζω έχει επίγνωση αυτών των κινδύνων και θα επικεντρωθεί στα ουσιώδη. Χαίρομαι που η πρωτοβουλία αυτή επιτέλους οργανώνεται ως διαρθρωτική απάντηση σε μια διαρθρωτική επίθεση των συνταγματικών μας αξιών, αρχών και θεμελίων της Ευρώπης. Όχι μόνο του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά έχουμε και το άρθρο 2 της Συνθήκης που προβλέπει τις θεμελιώδεις αξίες και τα βασικά θεμέλια της Ευρωπαϊκής Μεσένωσης. σα Σας ευχαριστώ θερμά για την στράτευσή σας την προσήλωσή σας στα θέματα αυτά και κάποια σημεία, κάποιες επικρίσεις θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη. Τα κριτικά σχόλια του Στεφάν και της Ζενεβιέβη είναι επίσης και εύλογα γιατί ε, ακόμη και η προάσπιση του καλού μερικές φορές μπορεί να μετατραπεί σε εξτρεμισμό κάτι που θα ήταν επικίνδυνο στην Ευρώπη και φαντάζομαι δεν αυτή η πρόθεσή σας. Πάντως είναι πολύ επίκαιρη η πρωτοβουλία σας και για τους καιρούς που διανύουμε. Και χαίρομαι που η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι μόνο απόδειξη ότι μια πρωτοβουλία των πολιτών μπορεί να βοηθήσει την οικοδόμηση της Ευρώπης, αλλά σας εύχομαι και επιτυχία για την πιστοποίηση, την επίστευση ε, την επαλήθευση των υπογραφών και ελπίζω να επαληθευτούν και οι εναπομείνασες υπογραφές και να επανέλθουμε μετά την επίσημη διαβίβαση των υπογραφών που θα κάνετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ακρόαση που θα γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν θα γίνει στο σημερινό κοινοβούλιο ή, το, ή στο επόμενο. Πάντω, ελπίζω να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Επίση, ε, θα ήθελα να σα ανακοινώσω ότι θέλουμε να διοργανώσουμε μια ειδική ιδιαίτερη συζήτηση στην Ολομέλεια του Μαΐου, όπως είπε και ο Στέφαν, μία εβδομάδα πριν τις εκλογές για το θέμα του αντισημιτισμού. Γιατί ο αντισημιτισμός είναι ένα επίσης ανερχόμενο φαινόμενο, δυστυχώς και πολύ επικίνδυνο εξτρεμιστικό φαινόμενο στην Ευρώπη. Θέλουμε να το πραγματευτούμε και να στείλουμε και εκεί ένα ηχηρό και ξεκάθαρο μήνυμα. Αυτά και θα περάσουμε τώρα στη δεύτερη συζήτηση του πρωινού. Όλα Λένερ, θα ήθελα να καλέσω τον πρόεδρο Μπερνασκόνη και την αντιπρόεδρο ε, της Γαλλικής Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Επιτροπής να έρθουν στο βήμα. Κύριε Πρόεδρε Μπερνασκόνη, κύριε Αντιπρόεδρε Κουβέρ, Αγαπητέ Πατρίκα, αγαπητή Καρόλ, σας εύχομαι πρώτα απ' όλα καλώς ήρθατε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως όταν σας υποδεχόμαστε εδώ στις Βρυξέλλες. Και είναι και ένας τρόπος έμπρακτος να σας ευχαριστήσουμε για την πολύ θερμή φιλοξενία που μας προσφέρατε πριν λίγους μήνες στο Παρίσι, στην, στο δικό σας ε, Οικονομικό, Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό Συμβούλιο που έχει τα ίδια αρχικά με την δική μας ε, Επιτροπή. Χαίρομαι για την αγαστή συνεργασία μας που είναι ε, παλιά βιώσιμη και σταθερή. Ο τη Αδεξιοπερή είχε πει ότι η πέτρα δεν έχει ελπίδα να γίνει τίποτα άλλο παρά πέτρα. Με τη συνεργασία, με τη συνεργασία της όμως με άλλες πέτρες μετατρέπεται σε ναό, σε τέμενος. Ας ε, συνεργαστούμε λοιπόν για να φτιάξουμε αυτό τον ευρωπαϊκό ναό, αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Πολλές ε, επιτυχίες είναι έμπρακτα παραδείγματα της συνεργασίας μας και συμμετέχουμε στις αιτήσει ε, συνεδριάσεις των εθνικών ΕΟΚΕ και αντίστοιχων φορέων στις δραστηριότητε του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Μάλιστα, πρόεδρος είναι ο Λόπο από την Πορτογαλία Έχουμε ε, θεματικές ε, συζητήσεις, ε, διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών και συνεργαζόμαστε σε πολλούς και διάφορους τομείς και θέλουμε να υπολογίζουμε σε εσά όπως έγινε στο παρελθόν για πολλά θέματα και κυρίως πρόσφατα στο θέμα της Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης. Και μάλιστα ο Γιώργο Δάση, ο προκάτοχό μου, είχε ξεκινήσει ευρύτατε διαβουλεύσει σε ολόκληρη την Ευρώπη, που στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία λόγω τη ε, αθρώση συμμετοχή και προσέλευση που είχαν. Επίση, ε, στι 18 Μαου του 2017 είχαμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση με εντυπωσιακά αποτελέσματα που συμπεριλήθησαν και στα δικά σας και στα δικά μας ψηφίσματα αλλά και στη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Πατρίκ, η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης θα ολοκληρωθεί στο άτυπο Συμβούλιο του Συμπίου στις 9 Μαΐου. Ε, με την ευκαιρία αυτή, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα πρέπει να δώσουν μια πολιτική απάντηση, απόκριση σε αυτή τη συζήτηση. Και μάλιστα το μήνυμα λίγο πριν τι ευρωεκλογέ ε, θα δώσει κάποιες ε, ε, αδρές γραμμές ε, για τις ε, αποφάσεις που θα ληφθούν στα Συμβούλια του τέλους Ιουνίου. Γιατί με βάση αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές θα δοθεί ο προσανατολισμός και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και από αυτήν την άποψη είχαμε και μια πολύ σημαντική γνωμοδότηση για το θέμα αυτό με τίτλο «Η Ευρώπη αφουγκράζεται τους πολίτες της». Ε, μάλιστα την γνωμοδότηση την εγκρίναμε χθε στην Ολομέλεια της ΕΟΚΕ και πολύ ευχαρίστω να σας διαβιβάσω την γνωμοδότηση αυτή. Εκεί περιλαμβάνουμε πολλά μηνύματα και επαναλαμβάνουμε την ανεπιφύλακτη υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών στο ευρωπαϊκό σχέδιο της αξίας και τα αποτελέσματά του. Η ΕΟΚΕ επιμένει στην ανάγκη να ε, χαράξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια παγκόσμια στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη το θεματολόγιο του 2030 για μια πραγματικά βιώσιμη Ευρώπη. Η βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να στηρίζεται σε μια ισορροπημένη στρατηγική που θα συμπεριλαμβάνει και την πρόκληση της ανταγωνιστικότητας αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία και την κοινωνική ένταξη. Επίσης, τονίζουμε την ανάγκη της προετοιμασίας ενός πραγματικού ψηφιακού μετασχηματισμού που θα επιτρέψει σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να παραμείνουν μοχλή δημιουργικότητας ε, σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Επίσης, ε, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε ως πρωταγωνιστές και όχι απλώς παρατηρητές τους πολίτες στην δημιουργία του μελλοντικού σχεδίου και φυσικά να ε, εμπλέξουμε πρώτα απ' όλα τους νέους σε όλα αυτά. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω μια άλλη σημαντική συμβολή της ΕΟΚΕ στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Είχαμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση με τίτλο «Η κοινωνία των πολιτών για την αναγέννηση» που έγινε στις 21 Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη Γαλλική ΕΟΚΕ και την Αντιπρόεδρο, την κυρία Καρόλ Κουβέρ, για τη συμμετοχή της στην συζήτηση με τους άλλους Προέδρους των αντίστοιχων Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων των κρατών μελών. Είχαμε πάνω από 400 συμμετέχοντες σε αυτή τη σημαντική, βαρισίμαντη εκδήλωση και 140 και δημοσιογράφους που κάλυψαν αυτή την εκδήλωση. Μάλιστα με την εκδήλωση αυτή στείλαμε ένα ηχηρό και απερίφραστο μήνυμα. Η Ευρωπαϊκή Κοινωνία των Πολιτών επιβεβαιώνει την αμέριστη υποστήριξή της στο ευρωπαϊκό σχέδιο με βάση ένα ισχυρό τρίπτυχο. Τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη νεολαία και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο. Ένα σχέδιο που θα είναι θεματοφύλακα των θεμελιωδών αξιών της, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, της κοινωνικής ένταξης, της αλληλεγγύης και της ανταγωνιστικότητας. Και με τις πρωτοβουλίες μας προσπαθήσαμε να κινητοποιήσουμε σε όλα τα επίπεδα την, ευρω... την κοινωνία των πολιτών εν ώψη των ευρωεκλογών. Και θεωρούμε ότι έχουν μεγάλη βαρύτητα οι επόμενες ευρωεκλογές και απαιτούν την επαγρύπνησή μας περισσότερο από, από ποτέ και τη δέσμευσή μας. Θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να συσπηρωθούμε για να έχουμε υψηλή προσέλευση στις εκλογές και μια ισχυρή και σαφή εντολή για να ενισχύσουμε τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ευρωπαϊκό σχέδιο για το μέλλον. Η ΕΟΚΕ συνεργάζεται με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα για να έχουμε ένα φιλόδοξο επικοινωνιακό σχέδιο που θα υπογραμμίζει τα επιτεύγματα και τα κεκτημένα της Ευρώπης, αλλά και τις αδυναμίες της και τις ανάγκες αλλαγής για να γίνει πιο αποδοτική και αποτελεσματική. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τον ευρωσκεπτισμό, και τον εξτρεμισμό και τον λαϊκισμό. Όλοι αυτοί χρησιμοποιούν οποιοδήποτε επιχείρημα για να μαυρώσουν ε, την εικόνα της Ευρώπης. Μερικοί δεν έχουν άλλη συνταγή παρά το να σπάσουν τα πάντα, να καταστρέψουν τα πάντα, να ρημάξουν τα πάντα. Εμείς όμως δίνουμε ένα εναλλακτικό όραμα ότι ε, η ενίσχυση του εθνικισμού και η απεμπόληση της μετανάστευσης δεν είναι η λύση για τα πάντα. Έχουμε περίπλοκα προβλήματα και χρειαζόμαστε πολυσύνθετες λύσεις. Θα πρέπει όμως να συσπηρωθούμε και να καταπολεμήσουμε το φόβο της μεταβαλλόμενης κοινωνίας. Ο φόβος αυτός μας στήχησε 60 ε, εκατομμύρια νεκρούς και 70 εκατομμύρια τραυματίες στην Ευρώπη τον περασμένο αιώνα. Θα πρέπει λοιπόν να διαφυλάξουμε την ειρήνη που τα τελευταία 60 χρόνια καταφέραμε να οικοδομήσουμε. Και γι' αυτό θα πρέπει να σφυριλατήσουμε πολλές συμμαχίες για να υλοποιήσουμε την αναγέννηση της Ευρώπης. Και γι' αυτό δημοσίως θα ήθελα να στηρίξω την επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος Μακρό, ανοιχτή επιστολή προς τους πολίτες στην Ευρώπη, που τον τίτλο είχε «Προς μια αναγέννηση της Ευρώπης». Δεν θα ε, ζητήσω copyright για το ότι με αντέγραψε ο πρόεδρος ε, Μακρό. Χαίρομαι γι' αυτό. Θα, συ... θα ολοκληρώσω με τα λόγια του φιλοσόφου Ζενζάκα Ρουσό. Ποτέ δεν είχαμε ένα τόσο ευγενές ε, και χρήσιμο όραμα όπως η αηφόρος και αιώνια ειρήνη μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Ευχαριστώ και σε ευχαριστώ Πατρίκ. Έχεις το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητέ Λουκά, αγαπητά μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, πριν εκφωνήσω την ομιλία μου, θα ήθελα να σας πω ότι με συγκινεί ιδιαίτερα η τιμή που μου κάνατε με την πρόσκλησή σας. Γιατί είχα δύο χρόνια να έρθω στην Επιτροπή σας και χαίρομαι ιδιαίτερος που θα έχουμε συζήτηση για τις ε, απόψεις μας σε μια ε, κέρια στιγμή και για το Γαλλικό Οικονομικό, Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι ένας από τους στόχους μας ε, έχει υλοποιηθεί, δηλαδή η σύσφυξη των δεσμών μεταξύ του δικού μας Συμβουλίου και της ΕΟΚΕ. Οι δεσμοί αυτοί διευκολύνουν ε, τη συνεργασία μας, που είναι και μια κοινότητα αξιών και αρχών και που εμπνέονται από μια μεγάλη αποφασιστικότητα. Και μάλιστα έχουμε μια προνομιακή σχέση εδώ και χρόνια με τους προέδρους σας. Αυτό ίσχυε και με τον Γιώργο Ντάση που θα ήθελα να χαιρετήσω γιατί ε, είχαμε μεγάλη συνεργασία μαζί του αλλά και με εσάς κύριε Γιάχερ και θα σας, ήθελα να σας καλέσω στο μέλλον, τον Απρίλιο στο Παρίσι για να έχουμε συζήτηση πάλι για το μέλλον της Ευρώπης, αντίστοιχη με αυτή που έχουμε και εδώ σήμερα. Λίγες εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογέ, κανένας δεν αμφιβάλλει ότι οι σκέψεις μας θα γίνουν ακουστές και παρά την κινδυνολογία θα θέλαμε να δώσουμε ένα μήνυμα βούλησης ανάκτησης και προάσπισης του ευρωπαϊκού ιδεώδους. Μπορεί να είναι ατελές αυτό το ευρωπαϊκό ιδανικό, αλλά η Ευρώπη είναι η μόνη πρωτότυπη πολιτική ε, λύση του 21ου αιώνα. Και δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική, γιατί οι υπόλοιπε με, μεγάλες δυνάμεις αναδιπλώνονται και κάτι, αυτό αλλάζει το σχετισμό των δυνάμεων. Οπότε έχουμε μια ένωση που δεν θέλουμε να αποδυναμωθεί, γιατί αν αποδυναμωθεί κάποια στιγμή θα εξαφανιστεί. Ε, εξού και μεγάλη έμπνευση που αντλήσαμε από την πρωτοβουλία αυτή των πολιτών με θέμα στο τον εξτρεμισμό που συζητήσατε πριν από λίγο. Το μέλλον της Ευρώπης σήμερα διακυβεύεται. Αφισβητείται και έσωθεν και έξωθεν από εθνικιστικές χήμερες όπως το Brexit και άλλους λαϊκισμούς που περισσότερο ε, έχουν ιδιοτέλεια παρά ειλικρίνεια. Και γι' αυτό θα πρέπει να αντιδράσουμε προβάλλοντας τα επιτεύγματα και τα πλανεκτήματα της Ευρώπης, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αντιδράσουμε και ε, πλησιάζουμε στην ανανέωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις ευρωεκλογέ. Να αντιδράσουμε, γιατί σίγουρα η Ευρώπη θα αναλάβει νέους στόχους, θα πρέπει να διορθώσει κάποια ε, λατώματά της, να βελτιώσει την εικόνα της, την επικοινωνία της, να έρθει πιο κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες να βελτιώσει αυτή την εγκύτητα, γιατί δεν προβάλλεται αρκετά. Θα πρέπει να δείξει ότι δεν είναι ούτε λόμπι, ούτε το παίγνιο των γραφειοκρατών, παρά την προσπάθεια που κάνουν οι λαϊκιστέ να την περιγράψουν έτσι, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για να εξυπηρετήσει του Ευρωπαίου πολίτε. Και επίση, για να επαναλάβω αυτά που είπατε όταν ήρθατε στο Παρίσι τον προηγούμενο Νοέμβριο, θα πρέπει η Ευρώπη να μάθει να αναπτύσσει ε, σχέδια που κοινοτοποιούν τους πολίτες, που τους ε, δημιουργούν ενθουσιασμό και να προτείνουμε τρόπους για να εξανθρωπίσουμε τη βιομηχανική επανάσταση, να λύσουμε την περιβαλλοντική κρίση που μας απειλεί όλου και πρώτα απ' όλα απειλεί του πλέον αδύναμους συμπολίτε μας. Και σίγουρα ε, δεν θα πρέπει να αποστασιοποιείται η οικονομία από την κοινωνία. Και μόνο με τέτοιες κοινέ λύσεις θα μπορέσουμε να ξανασεγινεύσουμε τους πολίτες και να τους επαναφέρουμε στο ευρωπαϊκό όραμα. Και νομίζω ότι είναι προφανές ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει ερήμη των πολιτών και χωρίς ε, την κοινωνία των πολιτών, χωρίς τους λαούς, χωρίς ε, αυτό το σημαντικό σώμα της Ευρώπης που είναι οι πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα δούμε και να επαναπροσανατολίσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε το σωστό ρόλο της Ευρώπης. Γιατί οι καιροί έχουν αλλάξει. Οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, ζητούν να ακουστεί ο λόγος τους και να εισακουστεί. Και εμείς οι ενδιάμεσοι φορείς, ε, ε, οι μεσάζοντες μεταξύ πολίτη και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή την θέληση. Δεν είμαστε απλοί παρατηρητές χωρίς δεσμευτικές απόψεις. Εμείς, και μπορεί να φαίνεται λαζονικό, είμαστε παράγοντες εξισορρόπησης και σοφίας και εμείς θα διευκολύνουμε με το διάλογο με τους πολίτες τη συνένεση και τι συμβαστικέ προτάσεις. Χρειάζεται μεταρρύθμιση και γι' αυτό η συμβολή μας ε, και η συνεισφορά μας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη γιατί είναι απαραίτητο εργαλείο για όποιον επιθυμεί την κοινωνική ειρήνη. Γνωρίζουμε τι εντάσει υπάρχουν ε, κυρίως στην πατρίδα μου το τελευταίο τετράμινο. Όλα αυτά είναι πολύ ενδεικτικές τάσεις ε, το αιτήματο της κοινωνίας των πολιτών και από τις αριστερές και από τις δεξιές παρατάξεις λόγω της έλλειψης ε, ε, διαλόγου και έλλειψη ευαισθησίας που μερικές φορές δείχνουν οι άρχουσες τάξεις. Μερικές φορές ε, γίνεται εκμετάλλευση της, των ταραχοποιών από την άκρα αριστερά και άκρα δεξιά σε όλα αυτά τα κοινωνικά κινήματα. Θα πρέπει να προλάβουμε λοιπόν τέτοιες χειραγωγήσεις και να περιορίσουμε τις διαστάσεις τους. Τα κίτρινα γυλάκια της Γαλλίας ε, δεν έφτασαν στο προσκήνιο ε, μόνο λόγω διαφορετικών ε, ιδεολογιών. Οι αγανακτισμένοι της Ισπανίας είχαν ξεκινήσει το κίνημα αυτό και ακολουθήθηκε από Έλληνες, Βρετανούς, Βέλγους και τώρα Γάλλους. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται από διοργανωτές ως διάβλος ε, διάδοσης μηνυμάτων και προκειμένου να αποφύγουμε ε, να έχουν ξεπεραστεί τελείως πλέον τα συστήματα προστασίας της δημοκρατίας μας πρέπει να εξελιχθούμε. Είχαμε και μία γνωμοδότηση ε, σχετικά με τον κατακαιρματισμό και την μετάβαση της γαλλικής κοινωνίας και τον αντίκτυπο επί της δημοκρατίας για μια έρευνα μέσω της καλύτερης ε, εκπροσώπησης, της καλύτερης συμμετοχικής δημοκρατίας, της καλύτερης συμμετοχής τελικά των πολιτών στις διαδικασίες των κοινών. Πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες ώστε να, συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες μας. Οι πολίτες πρέπει να είναι παρόντες στα κοινά, στη Βουλή, στη δημοκρατική διαδικασία. Εύχομαι ότι και η μελλοντική μεταρρύθμιση την οποία έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος Μακχόν θα είναι επιτυχής ώστε να έχουμε μια πιο συμμετοχική δημοκρατία. Εμείς δεν πρέπει να καθοδηγούμαστε αποκλειστικά από τα προεκλογικά ή μικροκομματικά συνθήματα. Και νομίζω ότι η Επιτροπή σας είναι η απόλυτη αντιστοίχηση, η απόλυτο συνεργάτης στην προσπάθειά μας αυτή. Όλα σε μια δημοκρατία είναι μια προσπάθεια εξέβρεση συμβαστικών λύσεων. Την περασμένη εβδομάδα, στην εβδομάδα για το περιβάλλον, έγινε αυτή η διαπίστωση θα μπορούσε κανείς να επιβιώσει ε, μέσα σε ένα δημοκρατικό σύστημα χωρίς συμβιβασμούς, χωρίς συμβαστικές προτάσεις και λύσεις. Όλα είναι θέμα λοιπόν ισορροπίας. Και φαίνεται να, να αναδύεται μια εξελικτική τάση. Και όλα αυτά πρέπει να οδηγήσουν στη μεταρρύθμιση του συμβουλευτικού Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού Συμβουλίου που είχε ήδη ανακοινώσει ο πρόεδρος Μακχόν από τον Ιούλιο του 2017. Σύντομα λοιπόν, ε, ποιοι είναι οι στόχοι αυτής της ε, προσπάθειας μεταρρύθμισης. Καταρχάς, να βελτιώσουμε τη διαδραστικότητα του Συμβουλίου αυτού με την κυβέρνηση, με το Εθνικό Κοινοβούλιο. για παράδειγμα με την υποβολή προτάσεων και έργων περιβαλλοντικού και κοινωνικού χαρακτήρα ώστε να αναδύονται οι προτάσεις που προέρχονται από την κοινωνία και να βρίσκουμε κοινέ κατευθυντήριες γραμμές. Να ενημερώνουμε καλύτερα τους πολίτες, να αποτρέπουμε τους κινδύνους κρίσεων. Δεύτερος στόχος είναι, όπως σας έλεγα, να βελτιώσουμε τη συμμετοχικότητα των πολιτών ε, στα δημοκρατικά κοινά. Να μπορούμε να διαβιβάζουμε τις πρωτοβουλίες των πολιτών χρησιμοποιώντας τα μέσα της ε, τεχνολογίας, της κοινωνίας, της πληροφορίας και να ενημερώνεται και να αναλαμβάνει δράση το Εθνικό Κοινοβούλιο επί των προτάσεων και πρωτοβουλίων αυτών. Εμείς μέσω αυτού του ε, συστήματος της διαδικασίας μεταρρύθμισης ευελπιστούμε, πιστεύουμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία της δημοκρατίας στη χώρα μας. Και αυτά έχουν σημασία και σε διεθνές επίπεδο μεταξύ των γαλλόφωνων χωρών για μια συνολικότερη προσπάθεια εκδημοκρατισμού των θεσμών και εκτός των συνόρων της Ευρώπης. Γιατί βλέπουμε ε, διεθνώς ε, τάσεις όπως στη Βραζιλία όπου ανεστάλλει η λειτουργία του αντίστοιχου, της αντίστοιχης κοινωνικής και οικονομικής επιτροπής. Εμείς πρέπει να ανοικοδομήσουμε γέφυρες με τους πολίτες όλων των χωρών ώστε οι ενώσεις, οι κοινωνικοί φορείς, οι οργανώσεις, οι πολίτες να επικοινωνούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και σκέφτομαι σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, ώστε να έχουμε μία αναθεμελίωση, όπως την ονομάζουμε εμείς, επανίδρυση δηλαδή, μια φιλοδοξία την οποία ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κύριε Πρόεδρε και με το σύνολο της ε, Επιτροπής σας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα επανέλθω σε αυτή τη σημαντική μεταρρύθμιση την θεσμική που έχετε ξεκινήσει και που ελπίζουμε ότι θα καρποφορήσει και θα ήθελα να ανοίξω τώρα τη συζήτηση με τα μέλη. Ο κύριος Σιβάσκου καταρχάς εκπροσωπώντας τη Ρουμανία για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω ρουμάνικα. Ε, πρόεδρε, από την χθεσινή ολομέλεια που είχαμε τοποθετηθεί για το μέλλον της Ευρώπης ε, και την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών, θα ήθελα να σας διαβιβάσω κάποιες από τις ιδέες που ομόφωνα εδέχθη η Ολομέλεια σχετικά με το ευρωπαϊκό όραμα και οικοδόμημα είχαμε τη συνάντηση του Σύμπιου και φυσικά όλη την περιπλοκότητα που απορρέει και την ασάφεια και την ανασφάλεια της διαδικασίας του Brexit. Προκειμένου να υπρασπιστούμε την κοινωνική δικαιοσύνη, την ελευθερία, την ισότητα και την διάκριση αρμοδοτήτων, δηλαδή τις αρχές και τις αξίες επί των οποίων έχει οικοδομηθεί η, Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίες δεν μπορεί να είναι διαπραγματεύσιμες, είναι αυτά στα οποία θα πρέπει να στηριχθεί το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η βιωσιμότητά του, η ισχύς του οικοδομήματος αυτού που πρέπει να βασίζεται σε κοινωνική σταθερότητα. Έχουμε σημειώσει σημαντικές εξελίξεις και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον μία από τις πολιτικά πιο σταθερές και πιο πλούσιες περιοχές στον κόσμο. Εξακολουθούμε όμως να έχουμε σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών σε επίπεδο κοινωνικής συνοχής. Πρέπει λοιπόν να συγκλίνουμε προς τα πάνω Πρέπει να έχουμε συνθήκες ε, εργασίας, συνθήκες διαβίωσης για τους πολίτες ε, βιώσιμες. Γιατί συχνά οι πολίτες θεωρούν ότι οι ωφέλειες από την συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχονται μόνο από τις κεντρικές κυβερνήσεις. Εξαρτάται το καλύτερο μέλλον από όλους τους πολίτες. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα επικοινωνίας που έχουμε στη διαθέσή μας. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα εθνικά, τις Εθνικές Κοινωνικές και Οικονομικές Επιτροπές, τις ΜΚΟ. Ο, ο Βικτό Ιγκό έλεγε ότι το μέλλον έχει πολλά ονόματα. Ας είμαστε θαραλέοι όπως μας προέτρινε να είμαστε ο Βικτόριο Ιγκό. Συγγνώμη, δεν ήθελα να ε, σας διακόψω την ώρα που παραθέτατε Ουγγό. Να δώσω τώρα το λόγο στον Γιάτσεκ Κράφτσικ, τον πρόεδρο της ε, πρώτης ομάδας των εργοδοτών από την Πολωνία, για τρία λεπτά παρακαλώ. Okay, good uh, morning everybody. Good morning, Mr. Ευχαριστώ, καλημέρα σε όλους, καλημέρα κύριε Πρόεδρε, εδώ είμαι. Είχαμε τη χαρά να συναντηθούμε και πριν από λίγους μήνες ε, στο Παρίσι. Σας καλωσορίζω στην ε, ΕΟΚΕ και χαίρομαι πολύ που βλέπω κάποιον που έχει κάποιο ε, υπόβαθρο κοινό με μας. Ξέρετε κι εσείς τι εκπροσωπούμε εμείς εδώ. Θέλω να είμαι πολύ σύντομος. Χθες η ομάδα μας η ομάδα των εργαδετών ενέκρινε μια διακήρυξη για μια ανοιχτή και συνεργατική Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να εργαστούμε για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ενότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μόνο μια ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί πραγματικά να μας υπερασπιστεί στο παγκόσμιο στερέωμα της αβεβαιότητας που αντιμετωπίζουμε πλέον. Έτσι θα μπορέσουμε να παράσχουμε ευημερία και ασφάλεια στους πολίτες μας. Επίσης πιστεύουμε ότι μια ενωμένη Ευρώπη μπορεί να είναι ισχυρή αλλά στην ποικιλομορφία της γιατί μόνο μέσω της συνεργασίας μπορούμε να δημιουργήσουμε εκείνους τους όρους ε, που θα μας επιτρέψουν να είμαστε αποτελεσματικοί και να έχουμε ε, επιρροή στο εξωτερικό. Φυσικά μπορούμε να Είμαστε περήφανοι ε, για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας και για την ευημερία. Αλλά για να υπερασπιστούμε αυτόν τον τρόπο ζωής θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον. Τι εννοούμε με αυτό. Θέλουμε να ε, μπορούμε τα έσοδα των επιχειρήσεων, ε, επιχειρήσεων να επιστρέφουν ε, στην παιδεία, στην υγεία, στην κοινωνία. Τα τρία στοιχεία που θέλουμε για το ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον είναι πρώτον, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το μέλλον. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε τις δεξιότητες, την καινοτομία και τις υποδομές, θα πρέπει να γίνουν κοινέ προσπάθειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη-μέλη. Ανοιχτέ αγορέ και ενσωμάτωση. Πρέπει να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά ε, να ενισχυθεί η ΟΝΕ και να ενισχυθεί το διεθνές εμπόριο. Επίσης χρειάζεται να υπάρξουν υποστηρικτικές συνθήκες για τους επενδυτές, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους επιχειρηματίες. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία πάνω στα οποία εμείς ε, βασίζουμε αυτό το νέο περιβάλλον που θέλουμε να χτιστεί, το ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις. Όλα αυτά θα πρέπει να συμβαδίσουν μαζί με τις αξίες. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να αμφισβητηθούν, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να, να αμφισβητηθούν οι αξίες Ευρώπης και μας ανησυχούν ε, τα αυταρχικά φαινόμενα που παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα. Πιστεύουμε ότι μια ανοιχτή κοινωνία και μια ε, ανοιχτή οικονομία θα ωφελήσουν όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Οι εργοδότες, οι επιχειρηματίες, οι άνθρωποι των επιχειρήσεων είναι και αυτοί πολίτες. και έχουμε πλέον το καθήκον να κινητοποιήσουμε τους πόρους μας. Οι ευρωεκλογέ είναι ευκαιρία και ευθύνη ταυτόχρονα. Είναι ώρα να δράσουμε. Κουλόν. Ε, και τώρα ο Κουλόν από το τμήμα Τένε. Τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Πατρίκ, πριν από λίγο μας είπες ότι είναι και η ώρα να ληφθεί υπόψη ο λόγος των φορέων μας, γιατί οι καιροί έχουν αλλάξει. Και δεν θέλουμε να είμαστε απλοί παρατηρητές της πολιτικής δράσης, με μόνο δικαίωμα να εκπονούμε μη δεσμευτικέ γνωμοδοτήσεις. Ναι, λοιπόν, πιστεύω κι εγώ ότι είναι και η ώρα να αρχίσει να λαμβάνεται υπόψη σοβαρά ο λόγος μας, λόγος θεσμικών οργάνων σαν τα δικά μας, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αν θέλουμε και εμείς να γίνουμε φορείς του μέλλοντος και συνελεύσει του μέλλοντος, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε το παρελθόν. Να θυμηθούμε τι δημιούργησε τη δύναμη, τον πλούτο των προτάσεων της ΕΟΚΕ. Το πλούτο, τη δύναμη τις προτάσεις ε, του, Ευρωπαϊκού, του Γαλλικού Οικονομικού, Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού Συμβουλίου και σε καμία περίπτωση αυτό το παρελθόν και όλες αυτές τις προτάσεις και την ισχύ θα πρέπει να τα ξεχνούν οι πολιτική μας. Όταν ο πρόεδρος Μπενασκόνη μας είπε ότι θα πρέπει να γίνουμε ένας φορέας ε, ε, και μια πλατφόρμα της κοινωνίας των πολιτών και οργανωτής κοινωνικών διαβουλεύσεων, μου θυμίσετε μία πρόσφατη συζήτηση που είχαμε στην ΕΟΚΕ για το τι μορφή θα πρέπει να λαμβάνουν οι δημόσιες διαβουλεύσεις και ποια θα πρέπει να είναι η συμμετοχή των κοινών θεσμικών οργάνων. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είμαστε οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Αλλά η αντιπροσωπευτικότητα δεν είναι η ίδια που ίσχυε στο παρελθόν. Σήμερα οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι η ψηφιακή οδός προέχει μερικές φορές της άμεση οδού, της αντιπροσωπευτικότητας και της ε, διαβούλευσης. Δεν μπορούμε βέβαια να καίμε μαζί με τα ξερά και τα χλωρά, αλλά δεν θα πρέπει να θυσιάσουμε την ουσιαστική διαβούλευση που κάνουμε εμείς μόνο προς το όφελος της αποκλειστικής ψηφιακής διαβούλευσης. Θα πρότεινα λοιπόν να ενισχύσουμε και να συσφίξουμε τους δεσμούς μας και να έχουμε συγκεκριμένες συζητήσεις για την ενισχυμένη συνεργασία των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Ε, και όσοι έχουν τέτοια βούληση και θέληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προετοιμάσουν από κοινού τις πραγματικές διαδικασίες διαβούλευσης, την πραγματική αντιπροσωπευτικότητα, την πραγματική εκπροσώπηση της κοινωνίας των πολιτών. Γιατί δεν α, θα, δεν θα μας λάβουν υπόψη. Ξέρουν οι Ιταλοί τι συμβαίνει με το Εθνικό του Συμβούλιο. Θα πρέπει να προλάβουμε αυτές τις εξελίξεις και όχι να είμαστε ουραγοί. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον Πατρίκ Μπερνασκόνη που πολύ τακτικά μας υποδέχεται στο μέγαρο ε, της περιοχής εκείνη στο Γενά και ελπίζω να συνεργαστούμε για να φτιάχνουμε από κοινού το οικοδόμημα. Ο Τζέιμ Μόρις τώρα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τη Βόρεια Ιρλανδία μάλιστα. Thank you very much. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό έχω, οπότε θα μιλήσω από καρδιάς. Είπατε ότι είμαι από τη Βόρεια Ιρλανδία. Είναι το επίκεντρο της καταιγίδα του Brexit η Βόρεια Ιρλανδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να φέρει την ειρήνη στην περιοχή από την οποία κατάγομαι εγώ. Το ίδιο μπορεί να, να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό που είπατε όμως είναι ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε πάνω απ' όλα είναι να εμπνεύσουμε τους νέους μας, να κινητοποιήσουμε την φαντασία τους, να τους δώσουμε λόγους και ελπίδα για το μέλλον. Αλλά το ίδιο και για τους εργαζόμενους μας, για τους ηλικιωμένου μας, για τα παιδιά μας. Πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να υπερβούμε αυτόν τον διχασμό που κινδυνεύει να ε, μας εκτροχιάσει και να καταστρέψει όλα όσα έχουμε κατακτήσει. Νομίζω ότι ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ένας δρόμος ηγετικός για την Ευρώπη ε, που θα μας δίνει ακριβώς τον λόγο για να ε, συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας στον κόσμο. Ευχαριστούμε, Τζέιν. Από τη Γαλλία, τους εργοδότες, έχει το λόγο εκπρόσωπος. Ευχαριστώ και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Πατρίκ, αγαπητέ Αντιπρόεδρε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως που σας υποδεχόμαστε εδώ σε αυτήν την αίθουσα του του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν μπορεί να, μην έχει το μεγαλείο του μεγάλου Ιένα αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία στην εκπόνηση της κοινοτική νομοθεσίας και του κοινοτικού προϋπολογισμού. Και πραγματικά έχουμε μεγάλη καινοτομία, ψηφιοποίηση, εξυγχρονισμό και προώθηση του ρόλου των γυναικών στο Γαλλικό Οικονομικό, Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό Συμβούλιο. Είναι αξιοσημείωτη και αξιοθαύμαστη συμβολή σας και μάλιστα εξυγχρονίζεται και τα μέσα της συμμετοχικής δημοκρατίας. Και αυτά όλα μας ενδιαφέρουν, γιατί έχουμε κοινό στόχο. Θα πρέπει να έρθουμε πιο κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες. Θα πρέπει να ε, προσανατολίσουμε καλύτερα στο μέλλον τι κοινοτικέ πολιτικέ και να το αντιληφθούν αυτό οι πολίτε. Το κάνετε εσεί στη Γαλλία και εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σίγουρα θα αλληλοδιδαχθούμε από τι εμπειρίε ε, και τι πολιτικέ μα για τα μέσα συμμετοχική δημοκρατία. Πάνελ πολιτών, όπω μα είπατε. Είχατε οργανώσει ένα παρόμοιο τέτοιο πάνελ πρόσφατα και εμεί το ίδιο στο παρελθόν με πολύ θετικά αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε με τέτοιες διοργανώσεις. Επίσης, επεξεργασία των αναφορών ή των ε, διαφόρων αιτήσεων των πολιτών. Ε, και εδώ θα μπορούσαμε να μιμηθούμε το παράδειγμα της Γαλλίας. Επίσης, έχουμε αναπτύξει νέες μορφές συμμετοχής, ε, με ευρύτερη συμμετοχή, με προσιτή ε, αυτή τη διαδικασία σε όλους τους πολίτες. Επίσης, ε, έχουμε οργανώσεις στις οποίες δεν καλούμε μόνο ομοειδεάτες. Θέλουμε αντιπαράθεση Θέλουμε γόνιμη συζήτηση με διάφορα επιχειρήματα ώστε να γίνει μια εκτενή συζήτηση για το ευρωπαϊκό σχέδιο. Οπότε μπορούμε να διδαχθούμε από τις κοινέ μας εμπειρίες και να κάνουμε μια τέτοια καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων. Και δεν θα πρέπει να σταματήσει αυτή η συνεργασία μετά τις ευρωεκλογέ, μετά τις 26 Μαΐου. Είναι ένα μακρόπνο έργο και όπως έλεγε και ο Σέντεξ Περί, η δημοκρατία θα πρέπει να είναι μια αδελφότητα η ΔΕΜΗ θα είναι μια φενάκι. Και νομίζω ότι και το Γαλλικό Συμβούλιο, το Οικονομικό, Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό, όπως και η Ευρωπαϊκή ΕΟΚΕ, μπορούν να γίνουν φορείς αδελφότητας, προτείνοντας και θεσπίζοντας νέες μορφές συμμετοχής και συνεργασίας για να διαφωτίσουμε αυτή τη συζήτηση και να την κάνουν κτήμα τους και οι πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς. Φυσικά έχουμε ε, περίπλοκες προκλήσεις, καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, κατανομή των πλεονεκτημάτων της ευημερία, ε, ποια είναι η κατάλληλη εμπορική πολιτική με συμμετοχή των πολιτών. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία και μπορείτε να υπολογίσετε στην δική μας υποστήριξη. Ευχαριστώ, Εμμανουέλ. Και τώρα, αν δεν με λένε, ε, ομάδα 2 Βέλγιο. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μπερνασκονή που ε, ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Ε, εκπροσωπεί ε, τις ενώσεις, τους φορείς αυτούς που είναι κρίσιμη σημασίας ώστε να διαβιβάσουν μελέτες, αναλύσεις, ιδέες ώστε να αναπτύξουμε συμφωνίες με τους κοινωνικούς εταίρους σε ένα σωστό επίπεδο και πολλαπλό επίπεδο. Συχνά έχουμε συστάσεις αναχώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του ε, εξαμήνου, αλλά πολύ συχνά, ακόμα πιο συχνά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγνοεί τις προτάσεις αυτές με άμεσο αντίκτυπο επί των μισθών, επί των θέσεων απασχόλησης, ε, των προγραμμάτων κατάρτισης ε, και της ε, βιώσιμης ε, περιβαλλοντικά και οικονομικά μετάβασης. Αυτά τελικώς έχουν έναν αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά και στην οικονομική κατάσταση και κοινωνική σύγκληση των χωρών και των πολιτών. Δεν πρέπει να εκπλησόμαστε νομίζω που έχουμε ψήφους διαμαρτυρίας υπέρ λαϊκιστικών κομμάτων, φαινόμενα διαμαρτυρίας όπως ε, τα κίτρινα γυλαίκα και δεν μιλώ για τους ε, καταστροφείς, μιλώ για αυτούς που πραγματικά αυθεντικά διαδηλώνουν. δεδομένων των πολύ φτωχών αποτελεσμάτων που έχουμε επιτύχει μέσω όλων αυτών των διαβουλεύσεων της διαδικασίας του κοινωνικού διαλόγου. Επομένως, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος κοινωνικού χάους όταν αγνοείται η δουλειά αυτών των ε, κοινωνικών οργανώσεων εκπροσώπησης. Αυτές οι διαδικασίες συμμετοχικής δημοκρατίας, τα δημοψηφίσματα μπορούν να διαδραματίσουν ένα κεντρικό ρόλο. Μπορούν να κινητοποιήσουν τη συμμετοχική δημοκρατία με τις ενώσεις, τις επαγγελματικές, τις ενώσεις εκπροσώπησης των εργαζομένων προκειμένου να αναπτύξουμε καλύτερα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Η άμεση δημοκρατία ή η εκπροσωπευτική δημοκρατία έχει και αυτή, καλώς κάνουμε και την ε, ευλογούμε, αλλά έχει και αυτή τα όρια της. Σε σχέση λοιπόν με το ευρύ κοινό, σε σχέση με τις αξιολογήσεις που πρέπει να κάνουμε ε, για τις πολιτικές που ασκούνται, για τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν πολιτικών προσανατολισμών κατευθύνσεων. Καθότι δεν έχουμε καρπούς στην κοινωνία. Τον λόγο για τον οποίο συγκεκριμένες κυβερνήσεις δεν παρακολουθούν τις προτάσεις από τις συμφωνίες που απορρέουν, ε, από τις συμφωνίες που έχουν γίνει μάλλον με τους κοινωνικούς εταίρους δεν, δεν χρειαζόμαστε, πιστεύετε, κάποιες, κάποια μέτρα που θα αποκαταστήσουν την αξιοπιστία των εκπροσωπευτικών αυτών οργανώσεων για να επιτύχουμε ένα κοινωνικό ε, όραμα, μια πραγματική κοινωνική πρόοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, αγαπητή Άννα. Χριστόφ Μπαλόν. Ομάδα 3. thank you very much. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την περσινή συνάντηση που είχατε με την πολωνική αντιπροσωπεία και την ε, επίσκεψη που έκανε η αντιπρόεδρός σας στη Βαρσοβία πέρσι. Ήταν πολύτιμη η συνεισφορά σας και για τη συζήτηση που διεξάγεται στην Πολωνία για το πώς μπορεί να βελτιωθεί στη χώρα ο κοινωνικός διάλογος και πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί και να δημιουργηθεί ένας νέος θεσμός προ αυτή την κατεύθυνση. Έχω ένα ερώτημα να σας απευθύνω που αφορά το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων στο οποίο αναφερθήκατε κι εσείς. Για μένα το σημαντικότερο ερώτημα είναι πώς γίνεται η συζήτηση στο Συμβούλιο σας σε σχέση με το κίνημα αυτό. Έχετε κάποιο μέλος του κινήματος που συμμετέχει στο Συμβούλιο σας. Κατά τη γνώμη σας, αποτελεί το κίνημα αυτό τμήμα της ε, κοινωνίας των πολιτών, της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών ή πρόκειται για ένα λαϊκιστικό κίνημα. Και το ερώτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η Γαλλία προφανώς και ανήκει στην καρδιά της Ευρώπης και επομένως ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία έχει πολύ μεγάλη σημασία για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπρέντα Κίνγκ από το Ηνωμένο Βασίλειο για τρία λεπτά από την ομάδα των εργοδοτών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την πραγματικά πολύ σημαντική ομιλία σας που μας ενέπνευσε και ως ε, Βρετανοί πραγματικά σας λέω ότι χρειαζόμαστε τέτοιες ε, ομιλίες. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ στο ζήτημα της Αφρικής και του εμπορίου. Ξέρετε ότι ο πρόεδρός σας έχει επισκεφτεί την Αφρική 16 φορές από τότε που εξελέγει. το ένα τρίτο αυτών των επισκέψεων έγινε σε αγγλόφωνες χώρες. Και ξέρετε ότι παλαιότερα είχαμε την τάση, την παράδοση, η Γαλλία να ασχολείται με τις γαλλόφωνες χώρες της Αφρικής και η Βρετανία στις αγγλόφωνες. Ε, όμως Η κυρία Μέη μάλιστα ε, πήγε και χόρεψε κάποια στιγμή κιόλας στην Αφρική ε, για να δείξει μια νέα στάση απέναντι στις χώρες. Εν πάση περιπτώσει, την προηγούμενη βδομάδα ο κύριος Μακρόν πήγε στην Κένια για την έναρξη του έργου 308 που είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που μπορεί να βοηθήσει και να ενισχύσει το εμπόριο ανάμεσα στην Αφρική, την Κένια, την Γαλλία και συνολικά την Ευρώπη. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι πώς μπορούν να συνεργαστούν οι δύο επιτροπές ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος όχι μόνο των Γάλλων εν προκειμένου αλλά και συνολικά ε, υπέρ όλων των Ευρωπαίων. Η Επιτροπή αυτή βεβαίως συμπεριλαμβάνει στους κόλπους της ε, την, τους εκπροσώπους της κοινωνίας των ε, πολιτών και στην Αφρική και στην, στην Ευρώπη κυρίως, αλλά πολύ συχνά έχουμε ε, εδώ ε, προσκεκλημένους και από την Αφρική, από την κοινωνία πολιτών των, ε, της Αφρικής. Θα γίνει και μια τέτοια εκδήλωση τον Ιούνιο που μας έρχεται. Εσείς ε, τι αποτέλεσμα θα προσδοκούσατε από τέτοιου είδους συναντήσεις που έχουμε. Ευχαριστώ κύριος ε, Γιώργος Ντάσης, ο προκάτηχός μου από την Ελλάδα γαλλόφιλος εδώ και πολλά χρόνια. Πώς το ξέρεις. Κάνουμε παρέδο και πολύ καιρό. Σε συναναστρέφουμε αρκετό καιρό. Ευχαριστώ Λούκα. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε Μπερνασκόνη. αγαπητέ Πατρίκ. Α, αγαπητή Καρόλ. Χαίρομαι ιδιαίτερος που σας βλέπω εδώ Είμαι πανευτυχής γιατί η συνεργασία μεταξύ ΑΟΚΕ και Γαλλικού Οικονομικού, Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού Συμβουλίου είναι παλιά. Ξεκίνησε και έλαβε χώρα και στη δική μου Προεδρία και είμαι περιχαρής που συνεχίζει αυτή τη συνεργασία και ο Λούκα. Και σας ευχαριστώ για την ομιλία σας που ήταν πολύ ε, χρήσιμη και παρόλο που έρχομαι από τον κόσμο των εργαζομένων και εσύ από τον κόσμο των εργοδοτών, θα μπορούσα κάλλιστα να προσυπογράψω όλα όσα είπες για την Ευρώπη. Για την Γαλλία θα τολμούσα να εμπλακώ. Σε ευχαριστώ απλώς και καταγράφω την πληροφορία που μας έδωσες. Άλλωστε, σήμερα, δεν ξέρω αν το αντιλήφθηκαν όλοι, υπάρχει μια γενική συνένεση και συνεννόηση για την ανάγκη να συνεχίσουμε να διαβιούμε σε αυτή την ειρηνική Ευρώπη. Είπε, αγαπητέ Πατρίκ ότι θα πρέπει να προασπίσουμε την μεγάλη ευρωπαϊκή ιδέα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνούμε. Θα πρέπει όμως να δούμε πώς θα την υπερασπίσουμε αυτή την ιδέα, αυτό το ιδεώδες. Και ήδη έδωσες κάποιες προτάσεις τις οποίες εστερνίζομαι. Σίγουρα θα πρέπει να αποσυνδέσουμε την οικονομία από την κοινωνία. Κάτι που δυστυχώς ε, ξεχνούν πολύ συχνά κάποιοι συνάδελφοι από την ομάδα εργοδοτών. Μερικές φορές, όχι πάντα. Επίση, είπε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει χωρί του λαού, ερήμην των λαών. Αυτό όντω ισχύει και είναι μια πραγματικότητα που τη γνωρίζουν όσοι έχουν διαβάσει την ευρωπαϊκή ιστορία, τουλάχιστον του περασμένου αιώνα. Πώ λοιπόν θα υπερασπίσουμε την ε, μεγάλη ευρωπαϊκή ιδέα. Καταρχήν θα πρέπει να ενημερώσουμε του νέου. Γιατί οι νέοι πιστεύουν ότι γεννήθηκαν στην ειρήνη και τη λαμβάνουν ως δεδομένη. Ε, θεωρούν ότι θα ζουν πάντα στην ειρήνη. Αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι δεδομένο, δεν είναι κεκτημένο. Θα πρέπει να προβάλλουμε τα επιτεύγματα τη ε, Ευρώπη που δεν είναι πάντα γνωστά, κυρίω τους νέου. Και επίση θα πρέπει να σημειώσουμε την πρόοδο που πρότεινε σε κάποια θέματα ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες, νέοι και λιγότερο νέοι, να συνεχίσουν να έχουν την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μοναδικό αγαθό για όλους. Τώρα, δεν θέλω να γίνω μακρονιστής για την πολιτική τάξη. Εγώ χαιρέτησα όλες τις πρωτοβουλίες του Προέδρου Μακρόν. Και όταν με ρώτησαν τη γνώμη μου, είχα πει τότε, είχα απαντήσει ότι το διάλογο το ξεκινήσαμε εμείς στην ΕΟΚΕ και εδώ και πολύ καιρό. Και η προάσπιση της ευρωπαϊκής ιδέας ε, είναι κάτι που συζητούμε εδώ και δεκάδες χρόνια στην Επιτροπή. Σε θέματα πολιτικής μετανάστευσης, ναι το ρολόι, ε, η Επιτροπή μας έλαβε πρωτοβουλίες πολύ πριν το Γάλλο πρόεδρο της Δημοκρατίας και πολύ πριν την εκλογή του. Ε, ο χρόνος δυστυχώς και το χρονόμετρο δεν μου επιτρέπει να μακρηγορήσω και να επεκταθώ. Πάντως πιστεύω ότι βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Λοιπόν, θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και με τα άλλα θεσμικά όργανα και τα άλλα συμβούλια για να, για να πείσουμε τους ηθήνοντες ότι χωρί να λάβουν υπόψη, αν δεν λάβουν υπόψη τα προβλήματα και τι προσδοκίε των Ευρωπαίων πολιτών, α ξεχάσουν την Ευρώπη. Και πολύ φοβούμαι ότι δεν θα χάσουμε μόνο την Ευρώπη, αλλά θα χάσουμε και την ειρήνη στην Ήπειρό μα, αν αγνοήσουμε τη βούληση των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιώργο. Ο Πίρκο Κοράναμαν από τη Φιλανδία τώρα για ένα λεπτό. Από την ομάδα 3. Κοίταξε, arvoisa Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, προσκεκλημένους μας, τους ομολόγους μας από την ε, αντίστοιχη Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή της Γαλλίας. Όταν μου είπατε ότι θα είχα ένα λεπτό στη διάθεσή μου, σκέφτηκα τι πραγματικά, σε, σε, σε ποια θέματα θα ήθελα να επικεντρωθώ. Η Ευρώπη μπορεί να έχει μέλλον μόνο αν τα πράγματα βαδίσουν σε σωστή κατεύθυνση. Και αυτό δεν αφορά μόνο την οικονομία, αφορά και τις πολιτικές στάσεις. Η πολιτική στάση του κάθε ανθρώπου λοιπόν διαμορφώνεται στην παιδική ηλικία και στην νεότητά του και που τον συνοδεύει η πολιτική αυτή στάση σε όλη του τη ζωή. Γι' αυτό θέλω να πω ότι η παιδική ηλικία, το περιβάλλον, η οικογένεια, αυτό είναι το σημαντικότερο για το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ Πύρκο, η κυρία Άγνες Σερ από την Ουγγαρία. Έχει και εκείνη ένα λεπτό στη διάθεσή της. Ε, γεια σας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας καλωσορίσω και εγώ κύριε, κύριε Μπερνασκόνη. Θέλω καταρχά να σας ε, συγχαρώ για την οικογενειακή πολιτική που ακολουθείτε, που υλοποιείτε στη Γαλλία. Είναι ο λόγο για τον οποίο δεν υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα στη Γαλλία. Μιλάμε σήμερα για το μέλλον τη Ευρώπη. Το μέλλον μα, δηλαδή. Είμαι απολύτω βέβαιη ότι το μέλλον τη Ευρώπη είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το μέλλον των παιδιών. Μίλησε και ο Πύρκο μόλι ε, πριν από λίγο για τη σημασία που έχουν τα παιδιά και οι μελλοντικέ ε, γενιές. Νομίζω ότι πραγματικά είναι σφάλμα από την πλευρά μας που ε, ασχολούμαστε τόσο πολύ σχεδόν αποκλειστικά με τους νέους και αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα τα παιδιά και τις οικογένειες. Γιατί η Ευρώπη είναι το σύνολο, η συντεταγμένη των ε, οικογενειών της, των πολιτισμών της. Ευχαριστώ πολύ. Και τελευταία παρέμβαση από τον κύριο Αρνό Σβάρτς από τη Γαλλία. Καλημέρα και ευχαριστώ όλους για τις ε, εισηγήσει τους ε, τους δύο προέδρους ε, σε επίπεδο ευρωπαϊκό και γαλλικό της Επιτροπής μας. αυτό που ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαίτερα από τις εισηγήσεις σας ε, ήταν, είναι η αναγκαιότητα να λάβουμε υπόψη μας ε, τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους αλλά σε συνδυασμό με τις προκλήσεις της κοινωνικής που αντιμετωπίζουμε με την άνοδο του λαϊκισμού, με την άνοδο των ανισοτήτων και με την ανάγκη να έχουμε μια βιώσιμη οικονομία. Η ανησυχία εκφράζεται από όλους και εδώ και στη Γαλλία. Βλέπουμε, θα έλεγα, και στις δικές σας τοποθετήσεις μια προοπτική για το μέλλον. Βλέπουμε την ανάγκη να συμμετάσχουν οι πολίτες στις εργασίες μας. Ο Μπεγνάχ μας θύμισε και την ανάγκη πειραματισμού με νέες τεχνολογίες, με νέες ε, μεθόδους διάδοσης των μηνυμάτων μας. Θα μπορούσαμε λοιπόν ίσως στο ε, πλαίσιο αυτό, βλέποντας όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους που διαδηλώνουν με ειρηνικό τρόπο, αλλά αποφασισμένοι, απαιτώντας ανταπόκριση, απαντήσεις, λύσεις, ίσως θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε νεαρούς ανθρώπους ε, να συμμετάσχουν στη δουλειά μας. Πώς θα μπορούσαμε να το πετύχουμε αυτό και ευρωπαϊκά και εθνικά. Ευχαριστούμε Αρνό. Ε, ολοκληρώσαμε με τον κατάλογο των ομιλητών. Αγαπητέ Πατρίκ, ε, μάλλον δύο ημέρες θα χρειαζόσουν για να απαντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτήσεις και προκλήσεις που ελέγχθησαν, που ακούσαμε. Δεν έχουμε δύο μέρες. Αν μείνεις στα δέκα λεπτά, ίσως να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε απλώς αυτήν την ετάπα, αυτό το βήμα αυτής της συζήτησης. Δεν νομίζω ότι ακούσαμε και τόσες πολλές ε, προκλήσεις, Πρόεδρε. Ε, εγώ είμαι δημοκράτης, ε, είμαι προϊόν μιας διαφορετικότητας που εδώ και κάποια χρόνια ίσως δεν ήταν τόσο προφανής από προέρχομαι από ιταλικές ρίζες, από δηλαδή μετανάστες που ήρθαν στη χώρα πριν από κάποια χρόνια. Αυτή η διαφορετικότητα πρέπει να προστατευθεί, αλλά πρέπει και να εξελιχθεί. Νομίζω ότι ε, αυτή η παράλληλη συνεργασία των φορέων μας είναι απολύτως απαραίτητη. Αναφέρεται ο πρόεδρος Μακχόν ε, ε, στην μετάβαση αυτή που μου φαίνεται ότι πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά έχοντας τώρα αναγνωρίσει τη σωστή κατεύθυνση εάν ε, ε, περιορίσουμε το πρόβλημα απλώς στα, στους φορείς τους εκπροσωπευτικούς δεν θα πετύχουμε τίποτα. Γιατί μπορεί να ανακύψουν άλλες τάσεις. Πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθούμε στους πολίτες. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα της τεχνολογίας που έχουμε στην διάθεσή μας. Δεν ξέρω αν στο μέλλον θα είναι οι πλατφόρμες, τα πάνελ ε, ή οτιδήποτε άλλο, η λαχνή, αλλά πρέπει να πειραματιστούμε. Πρέπει να πειραματιστούμε με τις κοινωνικές ε, μεθόδους εκπροσώπησης για να δούμε τι λειτουργεί καλύτερα και τι λειτουργεί χειρότερα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύνδεσμο. Γιατί εάν οι πολίτες μια μέρα αισθανθούν ότι πραγματικά υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος, ότι μπορούν να εκφράσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ότι έχουν ένα εργαλείο που τους επιτρέπει να μεταδώσουν, να εκφράσουν τη φωνή τους, να μεταδώσουν το, μήνυμά τους, θα μπορέσουμε να ενσαρκώσουμε ε, αυτήν, την, αυτό το σύνδεσμο που έχει χαθεί μεταξύ της πολιτικής ηγεσία και του κοινού. Αλλιώς θα έχουμε νέες τάσεις όπως αυτές που εκφράστηκαν στη Βραζιλία με την εκλογή της κυβέρνησης αυτής που είχαμε. οι χώρες εκείνες προσπαθούν να υποστηρίξουν δημοκρατικά συστήματα πρέπει να κατανοούν ότι πρέπει όλες οι ενώσεις, όλοι οι εκπροσωπευτικοί φορεί τους να έχουν τη δική της φωνή και να ακούγεται αυτή η φωνή. Και μια, μια κουβέντα για τους νέους ανθρώπους που είναι από τις πιο σημαντικές ανησυχίες μας. Τώρα εγώ βέβαια είμαι εξιντάρης και άνω. Πρέπει όμως να έχουμε τους νέους μαζί μας. Οι κοινωνικές και οι οικονομικές επιτροπές πρέπει να έχουν συμμετοχή από τους νέους ανθρώπους και στη δική μας περίπτωση συμμετέχουν και όχι μόνο στα θέματα που αφορούν άμεσα στην νεολαία, αλλά σε όλα τα θέματα που συζητούμε. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τις ανησυχίες τους, το όραμά τους. Και πρέπει πάνω απ' όλα να, να χρησιμοποιήσουμε αυτήν τη νέα τεχνολογία, τα νέα μέσα που χρησιμοποιούν οι νέοι. Για τις ε, διαδηλώσεις, για, τους, ε, για τα κέντρινα γυλαίκα, για τις διεκδικήσεις, ε, τις κοινωνικές, ε, τις ε, εδαφικές στη χώρα μας, τα βλέπαμε αυτά να έρχονται. Βλέπαμε ομάδες του πληθυσμού που αισθάνονταν απελπισμένοι, εγκαταλελειμμένοι. Όλοι αυτοί εκφράστηκαν με μια αμεσότητα για την ευζοία τους, για τα έσοδά τους, την έλλειψη δηλαδή εσόδων. Και μετά βέβαια ε, δυστυχώς όπως συμβαίνει πάρα πολύ συχνά όταν έχουμε τέτοιες άμεσες διαδηλώσεις από τον κόσμο ε, ισχωρούν στα κινήματα αυτά εξτρεμιστικές τάσεις που αυτές εκφράζονται με το δικό τους καταστροφικό τρόπο. Αν μα είχαν ακούσει πριν από τρία χρόνια που είχαμε υποβάλει μια γνωμοδότηση για τη συμφιλίωση της Γαλλία, τη συμφιλίωση της χώρας, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Γιατί έπρεπε να έχουν ληφθεί υπόψη μια σειρά από προβλήματα κοινωνικά που δεν ελήφθησαν. Αυτά λοιπόν τα, τα πηγαία κινήματα διαμαρτυρίας πολύ συχνά μετατρέπονται σε κύματα αγανάκτησης και τελικά μέχρι και βία περιστατικά. Για τον γαλλόφωνο κόσμο που σας έλεγα πριν, για τις χώρες της Αφρικής, ε, τις γαλλόφωνες αλλά και τις αγγλόφωνες, τις χώρες εν πάση τόσο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, έχουμε και εκεί φορείς κοινωνικής εκπροσώπησης και εκεί μπορούμε να βρούμε άξονες υποστήριξης της δημοκρατίας το ΣΥΖΑ, για παράδειγμα της Αφρικής. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτές τις κοινωνικές οργανώσεις των χωρών αυτών. Τώρα, πολύ σύντομα έχω φτάσει στο τέλος του χρονομέτρου ε, από τα λεπτά που μου έδωσε ο πρόεδρος. Ε, όταν με ρωτάτε τι περιμένω από τη σχέση μας, είναι περιμένω και ε, ευελπιστώ να μπορούμε να δρούμε συλλογικά από κοινού. Γιατί μόνο συλλογικά θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις και να βρούμε συνένεση στην κοινή γνώμη, στους πολίτες. Ε, εμείς ως Κοινωνική Επιτροπή Γαλλική και ως Ευρωπαϊκή θα πρέπει να ακούμε τους πολίτες μας. Να βρίσκουμε διαρκώς συνένεση όπως κάνουμε σε όλα τα επίπεδα εσωτερικά στη χώρα, σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε επαρχία, ώστε να έχουμε μια συλλογική προσπάθεια, μια συλλογική εκπροσώπηση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω ότι η παρουσία μου εδώ τέτοια μαρτυρία είναι. Πρέπει πιο συλλογικά να δρούμε και πιο συλλογικά να αποφασίζουμε. Χρειάζεται μια κοινή ομαδική προσπάθεια γιατί μόνο έτσι θα έχουμε τον σύνδεσμο μεταξύ των πολιτών και της ε, πολιτικής. Γιατί η έλλειψη εμπιστοσύνης, ε, η απώλεια εμπιστοσύνης στους πολίτες καμιά φορά είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Χρειαζόμαστε, ε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θερμά ευχαριστώ αγαπητέ Πατρίκ για την δέσμευσή σου, τη στράτευσή σου, τη συνεισφορά σου, τη συνεργασία σου. Τέσσερα συμπεράσματα θα ήθελα να αντλήσω. Πρώτον, δεν μπορούμε παρά να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς και με ιδιαίτερη προσοχή τη συζήτηση που θα γίνουν στη Γαλλία, που γίνονται στη Γαλλία, που προκλήθηκαν κάπως σκληρά στην αρχή με το πολιτικό κόσμο και μετά τη θεσμική μεταρρύθμιση του πρόεδρου Μακρόν και Ελπίζω με την ολοκλήρωση των συζητήσεων και των διαβουλεύσεων που έχετε να καταλήξετε σε μεταρρυθμίσεις ώστε να γίνει το Συμβούλιο σας ένα σώμα της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης με όλα τα συνεπαγόμενα. Ξέρω ότι κάτι τέτοιο φοβίζει τους γερουσιαστές, τους πολιτικούς, τους βουλευτές γιατί φοβούνται μήπως ε, λάβει υπερβολική εξουσία αυτό το τρίτο σώμα της Γαλλικής Βουλής αλλά πιστεύω ότι έχετε το κουράγιο και εσείς και ο πρόεδρος μακρόν για να ε, καταλήξατε σε τέτοιο συμπέρασμα μετά τη διεκπαιρέωση των συζητήσεων και των διαβουλεύσεών σας. ευχαριστώ που μου θύμισες κάτι που είχα ξεχάσει. Ένα ρητό του που είπε ότι η δημοκρατία μας, αν δεν καταφέρουν να γίνουν αδελφότητες, θα μετατραπούν σε φενάκι. Και για να κάνουμε κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τους ενδιάμεσους φορείς ε, σώματα σαν τα δικά μας, όχι γιατί είμαστε καλύτεροι οργανώσεις από άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Δεν έχουμε τίποτα καλύτερο, ούτε από πρακτική, ούτε από ηθική άποψη σε σχέση με άλλους ε, φορείς ή με τους πολιτικούς ή με άλλους θεσμούς. Απλώς εμείς ως διάμεσους φορέας έχουμε ένα σταγματικό στοιχείο, γιατί ε, αποκαλούσαμε ανέκαθεν την ΕΟΚΕ τον οίκο της κοινωνίας των πολιτών ή τον οίκο της ε, εργαζόμενης Ευρώπης. Είτε ο εργοδότης είναι κάποιος, είτε διευθυντής μιας τράπεζας, είτε διευθυντής συνεταιρισμού ή πρόεδρος μη κυβερνητική οργάνωσης ή αρχηγός συνδικαλιστικής οργάνωσης, κάθε μέρα χρειάζεται να εφεύρουμε λύσεις και οι λύσεις δεν πέφτουν από τον ουρανό ε, αναζητούμε τι καλύτερε λύσει, δεν θα κλείσει η επιχείρησή μα, η οργάνωσή μα, το συνδικάτο μα. Είμαστε υποχρεωμένοι να ε, κατασκευάζουμε συνεχώ και να δημιουργούμε συνεχώ. Γιατί έτσι ανανεώνομαστε και έτσι αυτά είναι τα στοιχεία τη αδελφότητα. Δεν χρειάζεται να έχουμε ένα υψηπετέ μεγάλο επίβολο σχέδιο. Ευτυχώ δεν έχουμε αυτή την ευθύνη, δεν είμαστε εμεί οι νομοθέτε, αλλά έχουμε μία δύναμη και θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Και περνάω στο τρίτο συμπέρασμα, στην τρίτη σκέψη. Θα πρέπει να αποφύγουμε ένα κίνδυνο. Γιατί αν ε, προσπίσουμε μόνο μια πάγια εικόνα των ενδιάμεσων φορέων, ίσως ε, μετατραπούμε σε ένα απολυθωμένο νεκροταφείο ή μουσείο. Μ' αρέσει η κεντρική πλατεία των Βρυξελών, αλλά μερικές φορές ε, αποτιμήσει και τη σημασία που είχαν οι συντεχνίε και κάποιοι τέτοιοι φορεί και από αυτό θα πρέπει να διδαχθούμε ώστε να παίξουμε έναν ανοιχτό ρόλο στη διαδικασία αυτή της ε, δημιουργία ανθεκτικότητα στον εξυγχρονισμό, στην καινοτομία και να διακινδυνεύσουμε κάποιε αλλαγέ και να μην προσπίζουμε μόνο τα πάγια και τα ε, κατεστημένα. Ε, και χαίρομαι για το έργο του κ. Μπερνασκόνη στο Γαλλικό Οικονομικό, Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό Συμβούλιο, γιατί είχε το θάρρο του πειραματισμού. Και μάλιστα μπήκατε σε αυτή την περίπλοκη διαδικασία των διαβουλεύσεων, ε, των άμεσων διαβουλεύσεων, των ψηφιακών διαβουλεύσεων, ακόμη και τη κλήρωση για τη συμμετοχή στι διαβουλεύσεις. Επίση, χρειάζεται διαδικασία συμβιβασμού και διαπραγμάτευση, αλλά χρειάζεται θάρρο για κάτι τέτοιο. Δεν θα πρέπει απλώς ε, να κρατήσουμε το ρόλο μας, να γίνουμε σαν την κεντρική πλατεία, κάτι πάγιο, κάτι μουσιακό. Θα πρέπει να γίνουμε ένας θεσμικός χώρος που ε, περιπείται αυτή τη διαδικασία διαχρονικά και όχι μόνο σε μια συγκεκριμένη στιγμή και την καλλιεργεί και τη φροντίζει. Και βέβαια είδαμε τους μπαχαλάκιδες που μπήκαν στα κίτρινα γυλαίκα και ήταν το ένα πέμπτο, αλλά πέντε φορές περισσότεροι ήταν όσοι, οι νέοι που κατέβηκαν ε, στα συλλαλητήρια για να προστατεύσουν το κλίμα. Α, αυτούς όμως δεν δόθηκε τόσο τέτοια δημοσιότητα. Επίσης, εξετάζεται μια θεσμική μεταρρύθμιση. Η Ευρώπη είχε μια πολύ σημαντική διέστηση που επιβεβαιώθηκε και από το δημοψήφισμα ε, και από τη, τη Βουλή, την Ευρωβουλή, η συνθήκη της Λισαβόνας που έχει τέσσερα άρθρα που προσδιορίζουν την ε, δημοκρατική διάρθρωση τη Ευρώπη. Το άρθρο 9 λέει ότι η Ευρώπη στηρίζεται στη δημοκρατία. Το άρθρο 10 λέει ότι το επίκεντρο τη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο χώρο που βρισκόμαστε. Το άρθρο 11 που προσδιορίζει την εντολή τη συμμετοχική δημοκρατία. που δεν ε, περιορίζεται μόνο στην διαβούλευση. Τρίτο εδάφιο είναι η διαβούλευση. Τα πρώτα δύο εδάφια του άρθρου 11 ζητούν τη συγκρότηση διαλόγου με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, με μόνιμο ε, και συγκροτημένο, διαρθρωμένο τρόπο. Δεν μιλά μόνο για διαβούλευση. Και το άρθρο 12 μιλά για το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων. Δεν είναι ότι ήταν μεθυσμένος ο πολίτης από το πολύ αλκοόλ όταν ε, ενέκρινε τη συνθήκη της Λισαβόνας και με δημοψηφίσματα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα άρθρα 10 11 και 12 μιλά για τη δημοκρατία που είναι η βάση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το άρθρο 11 λέει ότι ο θεματοφύλακας είναι, είναι ε, θεσμοί όπως η ΕΟΚΕ. Θα πρέπει λοιπόν ε, να, χρησιμοποιήσουμε αυτό το άρθρο και να αναβαθμίσουμε το θεσμικό μας ρόλο, να μην έχουμε μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα. Θα πρέπει να έχουμε το θάρρος για να καινοτομήσουμε και να βρεθούμε στο προσκήνιο όλων αυτών των διαβουλεύσεων και να πρωτοστατήσουμε σε αυτές. Και παρά την κόπωση, και η δική μας ε, Επιτροπή ε, καταφέρνει να είναι καινοτόμα. Και μάλιστα είχαμε με πολύ καλή πρωτοβουλία την Τρίτη ε, για τη συμμετοχή των νέων στην διαδικασία λήψη αποφάσεων. Την ε, διαδικασία ΓΕΣ που επινοήθηκε από την Αντιπρόεδρο της ΕΟΚΕ, την Ειρήνη Πάρη, την οποία και χαιρετίζω, και γίνεται με συμμετοχή όλων των, συμβου... σχολείων της Ευρώπης. Βέβαια, επιλέγεται ένα σχολείο αναχώρα. Ε, σήμερα το απόγευμα και αύριο θα έχουμε 105 ε, μαθητές από όλα τα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 5 -6, από 5-6 χώρες που έχουν ταξιακές διαπραγματεύσεις και εκπρόσωποι όλων αυτών των σχολείων θα συζητήσουν για τις ευρωεκλογέ και θα καταλήξουν σε συστάσεις και σε ένα ψήφισμα για να εκφράσουν αυτή τη θεσμική διάσταση. Και το κάνουμε εδώ και αρκετά χρόνια και νομίζω ότι είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη αυτή η θεσμική μας διάσταση. Ευχαριστώ και πάλι και είμαι ε, ευτυχής και υπερήφανος που συμμετέχουμε σε αυτόν τον αγώνα της ε, καινοτομία, όχι για να προασπίσουμε το θεσμικό μας όργανο και την ιστορία μας που ήταν λαμπρή και επιτυχής, αλλά για να οικοδομήσουμε το μέλλον ενός συγκεκριμένου χώρου της κοινωνίας των πολιτών που αυτή θα είναι η παρακαταθήκη που θα αφήσουμε. Και προσβλέπω στη θετική μας συνεργασία και σας ευχαριστώ και πάλι. I Περνάω τώρα τα καθήκοντά μου ως Προέδρου στην Μιλένα Αγγελόβα, για τις τρεις τελευταίες γνωμοδοτήσεις που θα συζητήσουμε και που πρέπει να εγκριθούν. Η Μιλένα λοιπόν θα προεδρεύσει τις διαδικασίες από εδώ και πέρα. Και θα το κάνει και καλύτερα από μένα γιατί είναι πιο αποτελεσματική και θα σας οδηγήσει και στη λήξη της ε, σημερινής ε, συνεδρίας της Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάμε στην ε, γνωμοδότηση εκπαίδευση για την Ευρωπαϊκή Ένωση της κυρίας Μπαμπραουσκιένε και του κυρίου Τραντίνα. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικό το σημείο στο οποίο είχαμε προβλέψει να συζητήσουμε τη γνωμοδότησή μας, γιατί ε, εν μέρη τουλάχιστον δίνει απάντηση η γνωμοδότησή μας στα προβλήματα και στα ερωτήματα που ανέκυψαν από τις ε, δύο προηγούμενες συζητήσεις που είχαμε. Υπάρχει ένα παράδοξο στην Ευρώπη. Αφενός γνωρίζουμε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για πάνω από μισό αιώνα κατάφερε να προσφέρει ευημερία, ασφάλεια, ειρήνη, αύξηση του επίπεδου, επίπεδου διαβίωσης και εργασίας των πολιτών της και αφετέρου ε, υπάρχει όλο και λιγότερη εμπιστοσύνη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στους εθνικούς θεσμούς. Αυξάνονται η τρομοκρατία, ο λαϊκισμός, ο εθνικισμός, υπάρχει παραπληροφόρηση, ψευδείς ειδήσει. Και όλα αυτά αποσκοπούν στην αποδυνάμωση των θεμελίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιος είπε ότι η πρωτοβουλία πολιτών αποτελεί μια θετική απάντηση, μια καλή απάντηση Κάποιοι διαφώνησαν με τη θέση αυτή. Εγώ θα έλεγα ότι δεν πρόκειται για τη λύση. Αυτό που πραγματικά πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι να ε, ε επικεντρωθούμε στα ριζικά αίτια των προβλήματων που αντιμετωπίζουμε. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται να δοθεί προσοχή στην εκπαίδευση. Η η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα πρέπει να έρθει πιο κοντά στους πολίτες και να ενισχύσει τις γνώσεις που έχουν οι πολίτες για τη σημασία και για τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δει κανεί το περσινό ευρωβαρόμετρο της Κομισιόν ε, ή τις, ε, τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών του 2014 θα δει ότι λιγότερο από ένα στους τρεις νέους συμμετείχαν στις εκλογές την προηγούμενη φορά. Το 28% μόλις των ανθρώπων 18 με έως 24 ετών συμμετείχαν στις τελευταίες ευρωεκλογές. Το Ευρωβαρόμετρο επίσης κατέδειξε ότι το 93% των Ευρωπαίων πολιτών ε, νιώθουν πολύ πιο κοντά στη χώρα τους και μόλις το 6% ε, ανέφεραν ή απάντησαν ότι θεωρούν ότι κατά κύριο λόγο η ταυτότητά τους είναι η ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη γνωμοδότησή μα, λοιπόν, περιλαμβάνουμε συστάσει και για το εθνικό και για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν μιλάμε για το ευρωπαϊκό επίπεδο, θεωρούμε ότι η ζωτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενίσχυση ε, της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Όταν δεν μιλάμε για την εκπαίδευση, δεν μιλάμε απλώς για την ε, αρχική εκπαίδευση ή την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μιλάμε για την εκπαίδευση στο σύνολό της, από μια ολιστική σκοπιά, ε, για τη διαβίου μάθηση, για την ατυπική μάθηση, ε, για την μάθηση για τους ηλικιωμένους. Και δεν μιλάμε στενά μόνο για την εκπαίδευση, μιλάμε και για την πληροφόρηση και την ενημέρωση των πολιτών. Γι' αυτό και ε, συστήνουμε τη δημιουργία θέσης επιτρόπου για την ενημέρωση και την εκπαίδευση. Γιατί θεωρούμε ότι αυτός είναι ένας κρίκος που λείπει αυτή τη στιγμή. Επίσης ζητούμε την αύξηση του προϋπολογισμού για το Εράσμους, γιατί θεωρούμε ότι η κινητικότητα στον τομέα της παιδείας από, για όλους τους πολίτες, από όποιο κοινωνικο-οικονομικό υποβαθρό και αν προέρχονται, είναι ζωτικής σημασίας ε, στοιχείο για το μέλλον της Ευρώπης. Έχω μόλις ένα λεπτό. Θα πω λοιπόν συνοψίζοντας ότι οι συστάσεις που περιλαμβάνουμε για το εθνικό και για το ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να μην είναι και ε, ε, να μην συμπεριλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που θα μπορούσε να, να συμπεριλάβει κανείς. Επικεντρωθήκαμε όμως στο να ε, καταρτήσουμε έναν κατάλογο όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένο με συγκεκριμένα μέτρα που συστήνουμε να ληφθούν και στο ευρωπαϊκό και στο εθνικό επίπεδο. Επίσης, περιλαμβάνουμε και κάποιες ρηξικέλευθες ε, ε, ιδέες, όπως για παράδειγμα ε, ε, να γίνει η 9η Μαΐου η ημερομηνία κατά την οποία θα μπορούσε να γίνει ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός όλων των δράσεων της, ε, της, επόμενης, χρονιές, της επόμενης χρονιάς ή ε, έχουμε και μια πρόταση για την ε, απονομή ενό βραβείου για εκείνους Ευρωπαίους πολίτες που προσφέρουν τα περισσότερα στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Ευχαριστώ πολύ. Πήρες δύο λεπτά από τον χρόνο που θα έδινα στον Πάβελ. Ε, Πάβελ παρακαλώ πολύ γρήγορα. Θα κάνω ό,τι μπορώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Αν ε, θα έπρεπε να συνοψίσω, το βασικό μου μήνυμα θα ήταν το εξής. Αντί για την, να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να ενισχύσουμε την μάθηση, γιατί είναι ολιστική, είναι διαβίου και ε, καλύπτει όλους τους τομείς της ζωής. Υπερβαίνει τις σχολικές αίθουσες και τις τάξεις και γι' αυτό αφορά όλες τις γενναίες και όχι μόνο τους νέους ανθρώπους. Όπως γνωρίζουμε, η εκπαίδευση ε, είναι, είναι μια διαδικασία που καλύπτει όλη τη ζωή και όλους τους τομείς. Με τρεις τρόπους. Τυπικά στα σχολεία, ατυπικά μέσω ε, οργανώσεων νεότητας και project και άτυπη ε, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ε, των συνομιλίκων κτλ. κτλ. Και θέλουμε όλοι και οι τρεις αυτές κατηγορίες, αυτά τα τρία είδη εκπαίδευσης να είναι αλληλοσυμπληρωματικά, ιδίω όσον αφορά την εκπαίδευση και την μάθηση γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκε ήδη ο αλφαβητισμός γύρω από τα μέσα ε, ενημέρωσης είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτεί κανείς από την παραπληροφόρηση που ε, είναι διάχυτη στις μέρες μας ε, γύρω μας. Δεν θέλω να πω για την, ε, δεν θέλω μιλήσω για την τυπική μάθηση και εκπαίδευση. Θέλω όμως να πω ότι στην μη τυπική εκπαίδευση βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορα project αυτή την περίοδο. Ξέρετε ότι υπάρχει μια, ένας συσχετισμός ανάμεσα στη διδασκαλία και την μάθηση και την απόκτηση εμπειριών γύρω από την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Όταν ε, κοιτάζω λοιπόν εδώ την αίθουσα και το κοινό που μας παρακολουθεί σήμερα, βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει για να μάθουν τις διαδικασίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να έχει κανείς απτές εμπειρίες για τις, εξι... για τις αξίες που διέπουν και διαπνέουν το έργο μας, για την ανάγκη συμβιβασμού ε, που μας χαρακτηρίζει πολλές φορές στο έργο μας. Ξέρω ότι εξάντλησα το χρόνο μου, κυρία Πρόεδρε, οπότε θέλω απλώ να ολοκληρώσω λέγοντας ότι είναι εξίσου σημαντική και η άτυπη μάθηση που προσφέρεται στους νέους ανθρώπους και μέσω του προγράμματος ε, «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή». Αν δε δείτε και το παράρτημα της γνωμοδότησης, το, ε, το, το οποίο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και μόνο. εκεί συμπεριλαμβάνουμε κάποια προγράμματα που θεωρούμε ότι μπορούσαν να μας εμπνεύσουν και για το μέλλον. Ακριβώς για να αποτυπώσουμε ακόμα καλύτερα αυτά που λέμε στη γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αγγλουνιάρ τώρα έχει το λόγο. Σας θέλω παρακαλώ όλους να τηρείτε το χρόνο αγόρευσης. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Είναι μια ιδεώδη στιγμή αυτή και πολύ επίκαιρη να μιλήσουμε για την εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το επίπεδο της γνώσης, ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δούμε, θα το διαπιστώσουμε στις επόμενες ευρωεκλογέ, γιατί θα είναι η στιγμή οι ευρωεκλογέ που θα επαληθεύσουμε τις μεθόδους ε, της προσέγγισης ε, των πολιτών, γιατί θα μιλήσουμε για τις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το μήνυμά μας θα είναι το μεγάλο κεκτημένο που δημιούργησε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ε, στις συζητήσεις φαίνεται ε, αν η ποιότητα της συζήτησης και η προσέλευση πληρούν τις προϋποθέσεις μας και αυτό θα δείξει αν ήταν καλό και το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αν όντως έγινε καλή ε, δεν υπήρξε καλή παιδεία. Γιατί αν η εκπαίδευση έχει μόνο ε, επιφανειακό χαρακτήρα και αν η προεκλογική εκστρατεία περιοριστεί σε κάποια στερεότυπα μόνο επιφανειακά για το ποια είναι τα υπέρ μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν φτάσει σε βάθος, δεν θα είναι ε, επαρκής. Και χαίρομαι που μιλήσατε για τον τρόπο που θα μπορούσαμε να τυποποιήσουμε την εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σίγουρα η επίσημη τυπική εκπαίδευση δεν είναι κοινοτική αρμοδιότητα, αλλά είναι σημαντικό η παιδεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει το αντικείμενο ενός ευρωπαϊκού σχεδίου. Και σε αυτό να προβάλλεται η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Τατιάνα και ο κύριος ε, Παύερ Ταραντίνα μίλησε για το πώς προσπαθούμε μέσω της επίσημης και τυπικής εκπαίδευσης προσπαθούμε να φτάσουμε και σε κάποιες φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης, άτυπης και θα πρέπει να έχουμε έναν κοινό χαρακτήρα και των, των τυπικών αυτών και της τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης όλα τα κράτη-μέλη. Μέχρι στιγμής είναι πολύ κατακαιρματισμένα αυτά τα σχέδια. Δεν υπάρχει ένα κοινό σχέδιο και χαίρομαι για την πρόταση Τατιάνα να έχουμε ένα πραγματικό εκπαιδευτικό προεδρείο, μια εκπαιδευτική επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να συντονίσουμε όλα αυτά τα μεμονωμένα σχέδια. Συμμετείχα στην ομάδα μελέτη και χαίρομαι ιδιαίτερω γι' αυτό. Δεν θα πρέπει να μείνει στα χαρτιά δυστυχώ αυτή η πρόταση, αλλά να κινητοποιήσει κάποιε δράσει ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Κοινωνία, αυτέ τι δράσει. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα και πάλι να σας θερμοπαρακαλέσω να μην υπερβαίνετε το χρόνο αγόρευσης για να μην φέρετε σε δύσκολη θέση να σας κόβω το μικρόφωνο. Ο κύριος Πετσίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η γνωμοδότηση συνδυάζεται και με την ε, δουλειά που κάναμε εχθές. Εγώ υποστηρίζω τη γνωμοδότηση αυτή και θα πρέπει να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο στο διάλογο μεταξύ μας η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εξαντλείται μόνο στα θέματα πολιτισμού και παιδείας. Πρέπει με, να το ενισχύσουμε με σύμβολα, με τους θεσμούς, ακόμα και με το στρατό, ε, με τις παραδόσεις. Ε, ε, στο παρελθόν ήμασταν πεπισμένοι ότι η συμμετοχή στην παράδοση αυτή θα είναι επαρκής, αλλά η αποτροπή του Ευρωπαϊκού Στρατού που μία συγκεκριμένη χώρα ε, ε, εθέλησε από πολύ παλαιά ε, οδήγησε σε μία έλλειψη ταυτότητας. Δεν φτάνει, επαναλαμβάνω, το εκπαιδευτικό σύστημα. Ένας Αμερικανός στρατιώτης λέει εγώ είμαι Μαρίν και εκπροσωπώ τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν δεν έχουμε αντίστοιχο αίσθημα ε, στην Ευρώπη, τότε οι εθνικισμοί, οι διάφοροι, ο γαλλικός, ο ιταλικός, ε, θα υπερνικίουν της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριος Μπάλης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν ζήτησα το λόγο για να ασκήσω κριτική στη γνωμοδότηση. Αντιθέτω, θέλω, θέλω να την υποστηρίξω. Έχω την αίσθηση ότι Υπάρχει όμως ένα θέμα το οποίο δεν έχουμε συζητήσει και δεν υπάρχει στην ε, γνωμοδότηση. Μιλώ για το e-learning, για την ηλεκτρονική μάθηση που έχει πολλές προοπτικές για το μέλλον και που πιθανότατα θα χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ακριβώς γιατί είναι αποτελεσματική σχετικά ε, φθηνή ε, και προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα και για τους νέους και για τους εργαζόμενους. Ίσως λοιπόν θα ήταν ε, καλό να συντάξουμε και μια γνωμοδότηση για την ηλεκτρονική μάθηση στην Ευρώπη γιατί θεωρώ ότι είναι μια μορφή που στο μέλλον πραγματικά θα μας αποφέρει πάρα πολλά ωφέλη. Very Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ιντζόβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μια ισχυρή γνωμοδότηση, πιστεύω, διότι σχετίζεται με τους βασικότερους άξονες αλλαγής στην Ευρώπη και ενδυνάμωσης κοινωνικής συνοχής. Μόνο η παιδεία μπορεί να μας βοηθήσει, έχει δίκιο η εισήγηση. Μιλούμε για κοινωνικές ισορροπίες και βλέπουμε και μια εστίαση στο πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερες ευκαιρίες για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Είναι ο καλύτερος τρόπος για την κοινωνική συμμετοχή και ένταξη. Σας ευχαριστώ κύριο Μουρτζιεύσκη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση για την γνωμοδότηση αυτή δεν θα πρέπει να αποκλεί αυτή την συμμετοχή σε αυτό το ρόλο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ε, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολλές φορές γίνονται κάποιες τοπικές ε, ενημερωτικές εκστρατείε ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιοποιούνται τα κοινοτικά κονδύλια στον πολιτισμό, στην παιδεία. Είναι πραγματικά η καθημερινή έκφραση του ευρωπαϊκού πατριωτισμού. η πρωτοβουλίες αυτές της τοπικής αυτοδιοίκησης και βλέπουμε καθημερινά στους πολωνικούς ε, δήμους και στις κοινότητες που είναι πάνω από 2.000 ε, στην Πολωνία. Θα πρέπει λοιπόν ε, να ενισχύσουμε την πληροφόρησή μας για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. 85% των κατοίκων της πολωνικής υπαίθρου είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στηρίζει τις ευρωπαϊκές αξίες. Δεν είναι αμεληταίο αυτό το στοιχείο. Σας ευχαριστώ κύριος Μπαλόν. Ευχαριστώ Μιλένα. Ε, ήμουν μέλος της ομάδας μελέτης και θα ήθελα να συγχαρώ ειλικρινά την εισηγήτρια και τον συνεισηγητή για το εξαιρετικό τους έργο. Και δεν το λέω μόνο για να μιλήσω. Δεν ε, ε, επιφανειακό το θέμα της γνωμοδότησης. Είναι πολύ περίπλοκο και πάρα πολύ σημαντικό και το αποτέλεσμα της γνωμοδότησης είναι αξιοθαύμαστο. Επίσης, ε, όταν συζητούμε την ε, ευρωπαϊκή ταυτότητα και τον ευρωπαϊκό πατριωτισμό, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η δημιουργία του δεν θα πρέπει να γίνεται από την κορυφή προς τα κάτω, αλλά από τη βάση προς την κορυφή. Αν έχουμε σχολεία ή με κυβερνητικέ οργανώσεις ή άλλους φορείς που προσφέρουν παιδεία και μάθηση, θα πρέπει να ξεκινήσουμε με την εξήγηση ότι σε αυτό το χωριό, σε αυτή την πόλη, ε, αυτό το χωριό και αυτή η πόλη είναι ευρωπαϊκά χωριά και πόλεις. Και γιατί? Ας κοιτάξουμε την ιστορία μιας περιφέρειας, μιας περιοχής, μιας πόλης, ενός δήμου, ενός χωριού ακόμη και να δώσουμε αυτή τη γνώση γιατί ένα χωριό είναι ευρωπαϊκό και γιατί μια πόλη είναι ευρωπαϊκή. Γιατί τα χωριά και οι πόλεις ήταν πάντα μέρη της Ευρώπης. Και τώρα έχουμε μια πολιτική δομή που μπορεί να μην είναι τέλεια. Θα μπορούσαμε να την αναπτύξουμε και να τη βελτιώσουμε, αλλά να ξεκινήσουμε ε, σε αυτή την ε, συμμετοχή μας στην οικοδόμηση, με τη συμμετοχή στις εκλογές και με τη συμμετοχή στην παιδεία. Είναι λοιπόν προφανές αυτό που θέλω να πω, ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα της παιδείας. Μπορούμε πρώτα να ξεκινήσουμε με την ενημέρωση για την Ευρώπη, για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να ξεκινήσουμε από τα στοιχειώδη. Ναι, ευχαριστώ, ξέρω, ξεπέρασα το χρόνο μου. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω γερμανικά. Νομίζω ότι μου είναι λίγο πιο εύκολο κάποιες φορές. Γνωρίζουμε όλοι, έχουμε όλοι πολύ λίγες γνώσεις σχετικά με την Ευρώπη, με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Αν πάει κανείς στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στους φίλους του, οι απαντήσεις ε, που θα πάρει είναι πολύ λίγες. Γι' αυτό και είμαι ευγνώμων απέναντι στην ε, ΕΟΚΕ για το γεγονός ότι μας έδωσε την ευκαιρία να εμβαθύνουμε σε αυτό το στρατηγική σημασίας ερώτημα και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να συνεισφέρουμε σε αυτό το, στη στρατηγική κατεύθυνση του μέλλοντος της Ευρώπης. Νομίζω ότι αν δεν το κάνουμε θα θέσουμε σε πολύ σοβαρό κίνδυνο το μέλλον της Ευρώπης. Κάποιοι ενδεχομένως ε, να ισχυριστούν ότι ε, ίσως ε, ήδη έχουμε χάσει πολύτιμο έδαφος και ότι θα μπορούσαμε διάφορες αρνητικές εξελίξεις να τις είχαμε αποφύγει αν είχαμε επενδύσει πιο έγκαιρα ε, και πιο πολλά στην εκπαίδευση. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω για αυτήν την ε, εξαιρετική γνωμοδότηση της Τατιάνα και του Πάβελ που συζητάμε σήμερα. Το έγγραφο πραγματικά από στρατηγική άποψης είναι άψογο παρά το γεγονός ότι χρειάστηκε στο τέλος ε, κάποια πράγματα να μπουν σε δεύτερη μοίρα γιατί προφανώς δεν γίνεται κανείς ε, να εντάξει όλη την κάμα των θεμάτων σε ένα ε, έγγραφο αυτού του είδους. Όπω για παράδειγμα η οικονομία. Πάντω, νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία ότι για την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια εύρωστη οικονομία και μια εύρωστη ανταγωνιστικότητα. Αποτελεί λοιπόν ε, το έγγραφο αυτό μια εξαιρετική βάση επί της οποίας μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο και να συνεχίσουμε να έχουμε και να χειριζόμαστε ως πρώτη προτεραιότητα την εκπαίδευση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Σίγκ. Um, <clears throat> uh, να σας συγχαρώ, να συγχαρώ μάλλον τον εισηγητή, τον συνεισηγητή και την ομάδα μελέτη για την εξαιρετική αυτή γνωμοδότηση. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση είναι κλειδί για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι βασικός λόγος της ύπαρξής της. Εγώ έχω παρακολουθήσει την καλή δουλειά που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις κοινότητές μας, στους δήμους μας. Έχουμε ανακοινώσεις σε όλους τους δήμους μας που λένε ότι τόσα χρήματα, τόσους πόρους συνεισέφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ε, με το Go Local, με μια τοπική δράση, θα είχαμε μια καλύτερη ίσως επιτυχία. γιατί οι βουλευτέ θυμούνται τι περιφέρειέ τους μόνο κάθε πέντε χρόνια που είναι εκλογέ. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα για να εκπαιδεύσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες και είναι ζωτική σημασία στην ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωση. Σα ευχαριστώ. Θα ξαναδώσω τώρα το λόγο στου συζητητέ ε, για δύο σύντομα σχόλια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, συμφωνώ πολύ με διάφορε από τι προτάσει. που ακούστηκαν εμείς είχαμε μια ομάδα μελέτης και ακολουθήσαμε φυσικά τις συστάσεις της. Ε, ο Σλάβορ βλέπω ήδη έφυγε, αλλά συμφωνώ ότι οι ευρωεκλογές ε, θα έχουν σημαντικά διδάγματα, όχι μόνο για το, σημείο, για το ποσοστό της συμμετοχής, αλλά και για τις επιλογές των πολιτών και για το πόσο ενδιαφέρονται, νοιάζονται για μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα στερεότυπα που έχουμε και την κατακαιρματισμένη πληροφορία και γνώση που υπάρχει. μιλούμε για την ευρωπαϊκή στρατηγική και για την εθνική στρατηγική και πρέπει να διατηρούμε υπόψη ότι η εκπαίδευση, τα θέματα της παιδείας είναι εθνική αρμοδιότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλώς έχει ένα συμπληρωματικό ρόλο εκεί. Δεν μπορεί να επιβάλλει εκπαιδευτικά προγράμματα στα κρατημέλη. Ε, κάποιος είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να καλύψουμε το τοπικό επίπεδο. Είναι αλήθεια. Νομίζω ότι πολλά μέλη μπορούν πράγματι να δραστηριοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο με πραγματικές δράσεις για τους πολίτες. Για, για το e-learning, ε, την προώθηση αυτής της κεντρικής πλατφόρμας και έχουμε διαφορετικές βεβαίως πλατφόρμες στο διαδίκτυο αλλά εμείς προσπαθούμε να αναπτύξουμε ένα μέσο διαδικτυακό με όλα τα εργαλεία που θα χρειάζονται οι διδάσκοντες. Ε, ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα απαντήσω στα τσεχικά. Για να απολαύσετε και λίγο την τσεχική γλώσσα. Καταρχήν σας ευχαριστώ για την υποστήριξη ε, ήταν μεγάλη χαρά τη συνεργασία μου με τα Τιάννα και τους άλλους εμπειρογνώμονε και τα πολύ δραστήρια μέλη της ομάδας μελέτης. Γιάτσε Κράφτσικ ε, ήταν εξαιρετικός ε, ως πρόεδρος της ομάδας και ευχαριστώ και τη Σαμπρίνα από τη Γραμματεία που επίσης μας βοήθησε. Και συμφωνώ ότι δεν αρκεί να μείνουν οι συστάσεις μας στα χαρτιά. Θα πρέπει να τις εφαρμόσουμε και εμπρά... Θα πρέπει να συνεννοηθούμε με την ομάδα επικοινωνίας για να δούμε πώς θα μεταβιβάσουμε καλύτερα το νόημα αυτής της γνωμοδότησης. Ο κύριος Πετσίνη είπε ότι τα σύμβολα έχουν σημασία. Συμφωνώ απόλυτα, γιατί τα σύμβολα προκαλούν αισθήματα και τα αισθήματα θα χαράξουν τις αξίες που χρειαζόμαστε στην εκστρατεία μας. Η Τατιάνα αναφέρθηκε και στο e-learning. Είναι σημαντικό να είμαστε δραστήριοι στο διαδίκτυο, να κάνουμε έντονη την παρουσία μας εκεί. Υπάρχει ένα site από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Τι κάνει η Ευρώπη για μένα». Πολύ χρήσιμος αυτός ο ιστότοπος. Η πρώτη τροπολογία μας αφορά το σημείο 6.1, είναι η τροπολογία 3 του Γκέρχατ Ρίμερ, γίνεται δεκτή. Είναι κανείς κατά. Όχι, οπότε εγκρίνεται η τροπολογία. Δεύτερη τροπολογία είναι η τροπολογία 2 για το 1-4 της συγγήτρια Μπαμπράου Σκένε και αυτή έχει γίνει δεκτή. Είναι κανει κατά. Όχι, οπότε εγκρίνεται και η τροπολογία 2. Τροπολογία 1 αφορά το 1-20 τη κυρία Oldfather. Έχει προταθεί ομω συμβαστική τροπολογία. Ποιο θα μα την παρουσιάσει. Είναι δύο οι τροπολογίε. Η τελευταία και η προτελευταία, δηλαδή τροπολογίε 1 και 4. Το συζητήσαμε με τους συντάκτες και με το συνεισηγητή προτείνουμε να συγχωνεύσουμε τις δύο τελευταίες τροπολογίες σε μια συμβαστική τροπολογία. Είναι αυτή που βλέπετε στην οθόνη. Ε, ξεκινάμε την πρώτη φράση. Σημειώνει τη φιλοδοξία που διατυπώθηκε στη διακήρυξη του Σούμαν, την οποία παρουσίασε ο Ρομπέρ Σούμαν στις 9 Μαΐου του 1950, σύμφωνα με την οποία η Ευρώπη δεν θα δημιουργηθεί διαμιάς, ούτε με βάση ένα συνολικό σχέδιο, αλλά θα οικοδομηθεί μέσα από συγκεκριμένα επιτεύγματα που καταρχάς θα δημιουργήσουν αλληλεγγύη. Η ΕΟΚΕ προτείνει η, μέρα της Ευρώπης 9 Μαΐου ή ακόμη και η διοργάνωση μιας ξεχωριστής Ευρωπαϊκής ημέρας εκπαίδευσης να επανεξεταστούν για το κατά πόσο θα μπορούσαν να εορτάζονται στα κράτη-μέλη και να χρησιμεύσουν ως αφετηρία για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα σχολεία και τις κοινότητες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλώς. Άρα καλύπτεται και την τροπολογία του Ξίστοφ Μπαλόν με τη συμβαστική τροπολογία. Έχει κάνει αντιρρήσει με τη συμβαστική πρόταση. Όχι, οπότε γίνεται δεκτή η συμβαστική τροπολογία και τώρα να ψηφίσουμε το σύνολο της γνωμοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία. Και σημειώνουμε μία επιπλέον ψήφο του συνεισηγητού. So I guess that we now can... Τέλος ψηφοφορίας. προσθέτουμε μία ψήφο. 164 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια στους συνεισηγητές. Και τώρα θα ζητήσω από την κυρία Χάινης να έρθει στο βήμα και να μας παρουσιάσει την γνωμοδότησή της υπαριθμών 874 για τις ψηφιακές δεξιότητες στον τομέα της υγείας και τον ψηφιακό γραμματισμό. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ε, μιλήσαμε εδώ και πάρα πολλή ώρα για την παραπληροφόρηση, την ψηφιοποίηση, για την εκπαίδευση και νομίζω ότι είναι εξαιρετικό το σημείο στο οποίο θα κληθούμε τώρα να συζητήσουμε τις ψηφιακές ε, δεξιότητες στον τομέα της υγείας. Ξέρουμε ότι η ιατρική όπως τη γνωρίζαμε έρχεται στο τέλος, έχει φτάσει στο τέλος της. Πλέον οι άνθρωποι πρέπει να είναι εκείνοι που θα γνωρίζουν τα πράγματα γύρω από την υγεία τους και θα πρέπει να έχουν και ψηφιακές δεξιότητες. Αυτό θα οδηγήσει ε, σε καλύτερο επίπεδο ποιότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών και από την σκοπιά των ασθενών βεβαίως που θα είναι πιο ενημερωμένοι αλλά και από τη σκοπιά των επαγγελματιών της υγείας. Οι ψηφιακές ε, δεξιότητες λοιπόν μπορούν ακριβώς να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που του προσφέρει η νέα ψηφιακή εποχή. Η ψηφιοποίηση αλλάζει όχι μόνο το πνεύμα αλλά και το σώμα των ανθρώπων. Οι ψηφιακές δυνατότητες λοιπόν ε, θα έχουν επιρροές και στον εγκέφαλό μας είτε το θέλουμε είτε όχι. Γι' αυτό και πρέπει να κοιτάξουμε την πραγματικότητα κατάματα, γιατί ο ψηφιακός κόσμος είναι ένας κόσμος φτιαγμένος από ανθρώπους, γι' αυτό και μπορεί να διαμορφωθεί με ευφυή τρόπο. Για την υγεία στην ψηφιακή εποχή, λοιπόν, ε, αυτό που προέχει είναι να καταστήσουμε τον ψηφιακό κόσμο φιλικό απέναντι στην ε, υγεία και να ενισχυθούν οι δεξιότητες στον τομέα της υγείας. Ο πολίτης λοιπόν θα πρέπει να παραμείνει το επίκεντρο της προσοχής των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Γι' αυτό και χρειάζεται μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τις ψηφιακές δεξιότητες στον τομέα της υγείας. Θα πρέπει και σε επίπεδο κρατών μελών να καταρτιστούν προγράμματα και σχέδια και να παρακολουθούνται αυτά άνθρωποι που έχουν ήδη γνώσεις γύρω από ψηφιακές δεξιότητες ε, μπορούν ήδη να παρακολουθούν καλύτερα την εξέλιξη της υγείας τους και αυτό αφορά ιδίως τους ηλικιωμένους. Η πρωτοβουλία λοιπόν ε, που αναλάβαμε ε, συμπεριλαμβάνει επιτυχή προγράμματα και έργα που έχουν υλοποιηθεί καλεί την Κομισιόν να συνεχιστούν αυτά τα προγράμματα, αλλά να ενισχυθούν και να συμπληρωθούν ώστε να μπορούν όλες οι πληθυσμιακές ομάδες και οι, τα άτομα με αναπηρίες και οι να μπορούν, ηλικιωμένοι να μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή. 70 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν, ε, είναι, είναι αναλφάβητοι. Ε, ακόμα περισσότεροι δεν ε, διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες κάτι που τους οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό, την ανεργία και τη φτώχεια. Δεξιότητες μπορεί κανείς να αποκτά σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, τυπικά ή και ατύπως, από την παιδική ηλικία. Οι θετικές επιπτώσεις μιας ποιοτικής ε, εκπαίδευσης είναι ε, πάρα πολύ ε, υψηλές. Η και ατυπως απο την παιδικη ηλικια οι θετικες επιπτωσεις μιας ποιοτικης ε εκπαιδευσης ειναι παρα πολυ ε υψηλες η οικογενεια το δημοτικό σχολείο είναι εκείνα που βάζουν τα θεμέλια για τη μελλοντική ικανότητα ενός ανθρώπου να αποκτά δεξιότητες και γνώσεις. Και εδώ εντάσσεται και η υγεία. Ένα έργο το οποίο εκτέλεσαν ασφαλιστικά ταμεία στη Γερμανία διαπίστωσε ότι πάνω από 55% των ενηλικιωμένων για το αν έχουν προβλήματα στο να κατατάσσουν και να κατανοούν τα προβλήματα της υγείας τους ε, απάντησε θετικά. Επίσης οι ίδιοι άνθρωποι απάντησαν ότι ε, η γραφή και η ανάγνωση δεν ανήκει στις δεξιότητες που κατέχουν ε, στον ε, βέλτιστο δυνατό βαθμό. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι ως Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή μπορούμε να συμβάλλουμε στην ευημερία των ανθρώπων ε, μέσω της της παροχής προς τους πολίτες της ε, δυνατότητας να κατανοούν τις πληροφορίες γύρω τους. Παλιά λέγαμε ένα μήλο την ημέρα κάνει το γιατρό πέρα. Τώρα πλέον μπορούμε να πούμε ότι μια εφαρμογή την ημέρα μπορεί να κάνει το γιατρό πέρα. Γι' αυτό και χρειάζεται μια ε, ολοκληρωμένη προσέγγιση όπως αυτή που επιλέξαμε μεταξύ των τμήματων της, Ευρωπα... της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Πρέπει να αναλυθούν σχετικές ε, πρωτοβουλίες. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα ε, σύνταξης της γνωμοδότησης, όλους τους ε, συναδέλφους και τη γραμματεία που μας υποστήριξε στεναρά. Σας ευχαριστώ ε, από ό,τι κατάλαβα έχουν υποβληθεί τρεις τροπολογίες και τις αποδέχεστε. Μάλιστα. Ε, δεν ξέρω αν έχει κάποιος αντίρρηση προς τις τροπολογίες αυτές. Ωραία. Άρα να σας ζητήσω να ψηφίσουμε τώρα για το σύνολο της γνωμοδότησης. Παρακαλώ. No, So now, uh... Πέρας της ψηφοφορίας. Α, όχι. Ε, ακόμα ψηφίζουν οι, οι συναδελφοί. Ωραία. Πέρας τώρα της ψηφοφορίας 153 υπέρ και 2 αποχές. Συγχαρητήρια. Θα ήθελα τώρα να καλέσω τον κύριο Κέρτις για την ΝΑΤ 754 προ ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για του ενδοκρινικού διαταράκτε. Ο κύριος Curtis. Okay, while we are waiting for Mr. Curtis. Λοιπόν, περιμένοντας τον κύριο Curtis, θα ήθελα να αναφερθώ και στα διάφορα υπό τα οποία θα ζητούσα από την Ολομέλεια να εγκρίνουμε για την αλλαγή Γιάσκους από Έκοσε Σοκ, Μάρτιν Σίκερ στο ΤΕΝ Άντερσεν αποχωρεί από την ΕΚΟ, Μπέντε Σόργεν Φράι, επίσης προς την ΕΚΟ, αν ακούσαμε καλά την Πρόεδρο. Η Ολομέλεια εγκρίνει θαύμα. Ο Μπράιαν έρχεται. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για τη μικρή μου καθυστέρηση. Πονούσε πλάτη μου από το, κάθισμα και έκανα μια βόλτα να χαλαρώσω λίγο την πλάτη μου. Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες είναι χημικές ουσίες που αλλοιώνουν τη λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος και επηρεάζουν αρνητικά στη ζωή των ανθρώπων και των ζώων. Μπορεί να είναι συνθετικές ουσίες ή φυσικές. Η έκθεση σε τέτοιες ε, ουσίες μπορεί να προέρχεται από πολλές ε, αιτίε. κατάλοιπα, λιπάσματα ή καταναλωτικά προϊόντα που ε, χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Το ενδοκρινικό σύστημα, όπω λέμε, είναι σύστημα γελιοφόρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χρησιμοποιείται ω επικοινωνιακό εργαλείο ε, και δίνει πληροφορίες ε, σε ιστούς, ε, όργανα, κύτταρα του σώματος. Μερικά παραδείγματα ενδοκρινικών διαταρακτών είναι οι δυσφενόλοι που καλεί για παιδιά, παραμπένες σε καλλιδικά ή σε πλαστικές ουσίες. Μάλιστα, η ανησυχία για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1990 και το 1999 η Ευρωπαϊκή Στρατηγική και ε, υιοθετήθηκε για τις, ε, για τις ουσίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που χρησιμοποιήθηκε για δράσεις ε, σε θέματα έρευνας και διεθνούς συνεργασίας. Και 20 χρόνια μετά την υιοθέτηση της στρατηγικής αυτής, η σχετική ανακοίνωση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως έλεγχος καταλληλότητας της κοινοτική νομοθεσίας. Έχουμε την επιστήμη για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και η πολιτική και η ρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά, ε, μάλλον η διεθνής ε, ε, νομοθεσία ακολουθεί την ευρωπαϊκή προσέγγιση. Για πρώτη φορά έχουμε μια τέτοια εγκάρσια εξέταση νομοθεσίας, στηρίζουμε, στηριζόμαστε σε επιστημονικά πορίσματα και που βασίζονται σε συνεχείς αξιολογήσεις των ουσιών αυτών. Επίση, θα έχουμε μία ετήσια ε, διάσκεψη των ενδιαφερομένων με συμμετοχή του ΟΣΑ κυρίως και άλλων διεθνών φορέων και θα ενθαρρύνουμε τα, κρα... θα ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν διάφορες ενημερωτικές ε, εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τους ε, ενδοκρινικούς διαταράκτες. Εμείς στηρίζουμε την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε να ενισχυθεί. Ε, οι σχετικές συστάσεις βρίσκονται στα, στο τμήμα για τα σχόλιά μας και ζητούν ε, πιο ευρείε διαβουλεύσεις με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών ε, γιατί η πρόταση σχετίζεται με την τρέχουσα νομοθεσία στα πλαίσια του 7ου ερευνητικού προγράμματο πλαισίου. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί με ρεαλιστικό σχέδιο δράση που θα έχει στόχου και προθεσμίε και θα εδράζεται στην εναρμονισμένη χρήση τη αρχή τη προφύλαξη. Τα σχόλια αυτά είναι ένα πολύ συνοπτικό, μια πολύ συνοπτική παρουσίαση των στόχων και με βάση τα επιστημονικά πορίσματα και τις γνωμοδοτήσεις αποφεύγουμε την εκτενή επιστημονική ανάλυση. Αν ε, επιθυμείτε κάτι τέτοιο, μια πιο διεξοδική ανάλυση επιστημονική, σας παραπέμπω στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως έχουμε μια πολύ, δύο πολύ ενδιαφέρουσες και δραστήριες ομάδες μελέτης και πολλές ε, Παρατηρήσει και προφορικέ και γραπτέ από τα κράτη-μέλη που λάβαμε υπόψη. Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα βοήθησε ιδιαίτερω. Ε, μας έστειλε εκπροσώπου στι και στι δύο ομάδες μελέτε και έπαιξε πολύ ενεργό ρόλο, κάτι που δεν ισχύει πάντα. Είχαμε ευρύτατε διαβουλεύσεις, Επίση είχαμε διαβουλεύσει με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τη βιομηχανία και από τους κορυφαίους εμπειρογνώμονε ε, της ε, παγκοσμίου παγκοσμίω εκτό των Ηνωμένων Πολιτών, τον καθηγητή Μαντοβάνη, και μα μίλησε για τα διάφορα στάδια και το τελευταίο, ε, ενημερώνοντάς μας για τις τελευταίες επιστημονικές εξέλιξεις και πορίσματα. Και ο David Sears, που είναι ε, χημικός, συνέταξε και πριν από μία δεκαετία μία έκθεση για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και συνέβαλε και αυτός στις εργασίες της ομάδας εργασίας που κατέληξε στην γνωμοδότηση. Όπως πολλές γνωμοδοτήσεις μας, ζητούμενο είναι η ισορροπία. Θέλουμε δηλαδή να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες της βιομηχανίας, των συνδικάτων και φυσικά και τις απόψεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και το γεγονός ότι η γνωμοδότηση πέρασε από το τμήμα χωρίς καμία αρνητική ψήφο και χωρί καν αποχέ, δηλαδή πέρασε επαμψηφή στην υποεπιτροπή, είναι απόδειξη μάλλον και μας ενθαρρύνει και εψυχώνει στο γεγονός ότι τελικά μάλλον καταφέραμε να βρούμε την ισορροπία. Ευχαριστώ θερμά τον εμπειρογνώμονά μου, την Επιτροπή, τη Γραμματεία και κυρίω τη Μόνικα που με βοήθησε ιδιαίτερος και φυσικά και τον καθηγητή Ματοβάνη που έπαιξε πολύ ενεργό ρόλο στην κατάρτιση αυτής της γνωμοδότησης. Σας ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ματιουλεβίτσιους. Ευχαριστώ πρόεδρε να συγχαρώ τον εισηγητή για εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά έκανε και ο ίδιος και ο εμπειρογνώμονάς του. Εγώ είχα την τύχη να είμαι στην ομάδα μελέτης. Είχαμε πραγματικά μια συζήτηση ψηλού επίπεδου και ποιοτική. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για την ευρύτερη κοινωνία. Ε, ε, ε, βλέπουμε τους διαταράκτες καθημερινή μας ζωή, στα τρόφιμά μας, ε, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να γνωρίζουμε τα θέματα αυτά. Εγώ χαιρετίζω την ε, δική σας πρόταση να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερη χρηματοδότηση για την έρευνα και ανάπτυξη νέων μέσων και εξερεύνησης των ενδείξεων του κατά πόσο έχουμε ε, επιμολυντές και κατά πόσον θα πρέπει να έχουμε μια αρχή προφύλαξης. Ε, όλες οι πράξεις μας πρέπει να έχουν επιστημονικές ενδείξεις και συμβουλές Βεβαίως παράλληλα είμαστε όλοι καταναλωτές και είμαστε όλοι γονείς. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει μια κατάλληλη στρατηγική, ιδιαίτερα με κρούσματα που μπορούν να πολλαπλασιαστούν απότομα και έτσι να πολλαπλασιάσουν τον αντίκτυπό τους. Ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή για την εξαιρετική του δουλειά και θα ήθελα και πάλι να αναφερθώ στην ποιότητα των γνωμοδοτήσεων του Βρετανού συναδέλφου που την εκτιμούμε και ελπίζουμε να τον έχουμε μαζί μας και, και στο μέλλον. Ε, σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Ράουνεμα. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για τη γνωμοδότησή του. Αρχικώς πρέπει να σας πω ότι είχα κάποιες αμφιβολίες, ήμουν κάπως επιφυλακτική για το τι θα μπορούσαμε να πούμε για αυτό το θέμα. Όμως ε, διαπιστώνω ότι το κείμενο τελικά είναι ισορροπημένο, βασίζεται σε τεκμήρια και σε στοιχεία και ε, αποσκοπεί στο να αναδειχθεί αυτό το πρόβλημα των ενδοκρινικών διαταρακτών τα οποία μεταφέρονται στον ανθρώπινο οργανισμό και μέσω των τροφίμων και μέσω των φυτοφαρμάκων. Και θεωρώ ότι πραγματικά πρέπει να υπάρξει σαφήνεια και διαφάνεια γύρω από αυτό το θέμα. Αν υπάρχουν αμφιβολίες πρέπει οι έρευνες να συνεχιστούν ώστε να μπορέσουμε συνολικά να διαμορφώσουμε μια σαφή εικόνα και να μπορέσει αναλόγως να δράσει και ο κλάδος των τροφίμων και των φυτοφαρμάκων. Γιατί αυτό που διακυβεύεται είναι πραγματικά η ζωή των ανθρώπων. Πρέπει λοιπόν να γίνουν έρευνες, χρειάζεται προφανώς στην κατεύθυνση αυτή να θεσπιστούν και συγκεκριμένες νομικές ρυθμίσεις με σκοπό ε, την προστασία των καταναλωτών, των επιχειρήσεων αλλά και των γεωργών που χρησιμοποιούν ε, τα φυτοφάρμακα αυτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριος Ρεάλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ζήτησα το λόγο ως πρόεδρος ε, του τμήματος ΝΑΤ. Ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά τον ε, συνάδελφο Brian Curtis για την εξαιρετική δουλειά και πολύ ισορροπημένη δουλειά. αλλά σκέφτομαι και τον καθηγητή Μαντοβάνη, ε, την κυρία Πόλιγκα, που όλοι έχουν ιδιαίτερη εμπειρογνωμοσύνη σε αυτήν τη θεματική και πολύ ε, καλά έκανε και τους επέλεξε. Εγώ θεωρώ ότι ο Μπράιαν ε, υπήρξε επίσης εξαιρετικός διότι πρόκειται για ένα θέμα δύσκολο, περίπλοκο, αλλά παρόλα αυτά συνδύασε τις πηγές και τις λύσεις που μπορούμε να βρούμε εδώ με μια προβληματική σε επίπεδο δημόσιας υγείας, έρευνας και ανάπτυξης και βιομηχανικής ανάπτυξης και συνεργασίας με τρίτες χώρες. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά θετικά. Η προσέγγιση του Μπράιαν βασίστηκε στην παρούσα ε, κατάσταση της ε, γνώσεως προσπαθώντας να αποφύγει αντιφατικά σημεία ή συγκρούσεις επί του θέματος των, θέματος των διαταράκτων που θα μπορούσαν να, είναι, να έχουν αποσταθεροποιήσει την γνωμοδότηση. Τον ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ κυρίως. Ντούφι. Ο κύριο Ντούφι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ ήμουν μέλος τη ομάδα μελέτη. Και πρέπει να πω ότι η δουλειά του Μπράιαν και του Προέδρου της ομάδας μελέτης ήταν πραγματικά εξαιρετική. Πρόκειται για ένα επιστημονικό πρόβλημα, πολύ συγκεκριμένο και δεν μπορούμε να το αγνοούμε. έχουμε ένα σύστημα ορμονών στο σώμα και αθένων που ελέγχουν όλες τις οργανικές μας λειτουργίες. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι κάποια από τα στοιχεία χαρακτηριστικά αυτά συνδέονται με τη διατροφή μας, δηλαδή εισέρχονται στο σώμα μας μέσω της διατροφής. η γνωμοδότηση αυτή νομίζω ότι ε, φτάνει σε θέματα που είναι πολύ μακριά από αυτά που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε τώρα και στα οποία δεν μπορώ να αναφερθώ, αλλά θα ήθελα απλώς να πω ότι δεν πρέπει να περιζόμαστε σε μία και μόλι γνωμοδότηση. Ήθελα να ζητήσω λοιπόν από την ε, Επιτροπή μας, από την ΕΟΚΕ, να δημιουργήσει μία μόνιμη ομάδα μελέτης των θεμάτων αυτών για να έχουμε τακτική ενημέρωση κάθε χρόνο σχετικά με τις αλλαγές και τις τάσει του συστήματος, διότι όλα αυτά σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα. Και ορισμένες τάσεις μπορούν να, να κινηθούν πολύ ταχύτερα από μας και να μην προλάβουμε με να τις παρακολουθήσουμε. Νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντικό θέμα όσο και η κλιματική αλλαγή για όλες μας τις χώρες. Ευχαριστώ τον Μπράιν, τον Βλαντίμιρ και όλους τους υπόλοιπους ε, της ομάδας μελέτης θα καταλάβουμε στο μέλλον πόσο σημαντικά είναι τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πιλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή μας για την εξαιρετική του γνωμοδότηση. Όπως είπα και προλαλήσαντε, το θέμα είναι περίπλοκο. Ε, εγώ το αντιμετώπισα τα τελευταία 20-25 χρόνια ε, στον κλάδο και φυσικά θα πρέπει να έχουμε μονίμως παγρύπνηση και εγρήγορση για το σημείο αυτό. Χαίρομαι εγώ, μίλησε για τα ανθυγιεινά προϊόντα από τρίτες χώρες, γιατί πέραν της επιστηστικής ασφάλειας ε, θα πρέπει να προσέχουμε τα εισαγόμενα προϊόντα που δεν είναι τόσο ασφαλή με τα δικά μας. Έχουμε πολλά συναρπαστικά προϊόντα που έρχονται πολλές φορές από την Αλοδαπή, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις και να είναι γεμάτα με ενδοκρινικούς διαταράκτες. Ευχαριστώ που το επισημάνατε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο Προελή σα μίλησε για τη διασύνδεση του θέματο αυτού με τι κλιματικέ αλλαγέ. Α μην ξεχνούμε όμω και του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη. 169 169 στόχοι δεν περιλαμβάνουν ίσως ενδοκρινικούς διαταράκτες, αλλά θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, γιατί είναι κλάδος που θα πρέπει να μας απασχολεί και να είμαστε σε επαγρύπνηση, όπως είπα. Ευχαριστώ τώρα ο λόγος τον κύριο Κέρτης για να απαντήσει στα σχόλια. Ευχαριστώ. Και τα αποκοκκινίζω με τόσες φιλοφρονήσεις ε, και κομπλιμέντα για την γνωμοδότησή μου. Όπως είπε και κάποιος όμως προλαλήσεις, είχα τόσο μεγάλη βοήθεια, τόσο ανεκτήμητη ε, βοήθεια και στην ομάδα εργασίας είχαμε πολύ καλή θέληση. Γνωρίζαμε πόσο σοβαρό είναι το θέμα, την ανάγκη να καταλήξουμε σε συμβασμούς και αυτή η συνειδητοποίηση μας διευκόλυνε πάρα πολύ. Και ο ε, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ομάδα εργασία και πολύ σωστά είπε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη χρηματοδότηση, περισσότερα κονδύλια και φυσικά την αρχή της προφύλαξης που θα πρέπει να εφαρμόζεται. Και είπαμε, εκτός από την αρχή της προφύλαξης, ε, ε, το plausibly, που κατά πάσα πιθανότητα έχουν ενδοκρινικούς διαταράκτες. Μερικές φορές ε, μπορεί να λέμε ότι και τα αντισυλληπτικά έχουν τέτοιους ενδοκρινικούς ε, διαταράκτες, αλλά δεν υπάρχουν ε, πορίσματα που να το επιβεβαιώνουν. Θέλουμε λοιπόν την αρχή της προφύλαξης κάποια στιγμή θεωρούσαμε ότι ο αμίαντος ήταν ακίνδυνος. Κανένα δεν θεωρούσε ότι υπήρχε πρόβλημα με τον αμίαντο. Μετά ανέκυψαν κάποιες αμφιβολίες. Αν τότε είχαμε την αρχή της προφύλαξης, θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε τον κίνδυνο και να σώσουμε χιλιάδες ανθρώπινες ζωές ε, που χάθηκαν εξαιτία αυτού του προβλήματο. Επίση, ε, ο Πέρκ ε, μίλησε για την βιομηχανία παραγωγή τροφίμων και τη γεωργία. Και εκεί θα πρέπει να επανέλθουμε στην ισορροπία, να σταθμίσουμε τους κινδύνους και να εξασφαλίσουμε μία εύρωστη βιομηχανία και ανθούσα. Και αυτό είναι σημαντικό. Επίσης, ο Μαουρίτσιο, ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας, μίλησε για τα εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες. Το ίδιο ανέφερε και ο Τζόναθαν Πιλ. Και εκεί θα πρέπει να επαγρύπνουμε συνεχώς για τα θέματα αυτά. Και επίση ε, άλλο συνάδελφο ο Μπόμ που έπαιξε ενεργό ρόλο στην ομάδα εργασία και μα κράτησε επικεντρωμένου και εστιασμένου σε πολύ σημαντικά θέματα για να μην μεροληπτήσουμε προ τη μία ή την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω αν χρειάζεται μόνιμη ομάδα εργασία. Πάντω σίγουρα το θέμα χρειάζεται μόνιμη επίβλεψη και προσοχή ε, μόνιμης γιατί σίγουρα αυτή δεν θα είναι η τελευταία γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Και το σχόλιο του Τζόναθαν για τη βιώσιμη παραγωγή, για την ε, ε, επαγρύπνηση που χρειάζεται, θέμα που ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι. Έχω συντάξει αρκετέ γνωμοδοτήσει. Αυτή θα είναι η τελευταία μου στην ΕΟΚΕ, εκτό και συμβεί κάτι. Ποιο ξέρει τι θα συμβεί στην πατρίδα μου. Πολύ φοβάμαι όμω ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτή θα είναι και η τελευταία μου γνωμοδότηση στην ΕΟΚΕ. Στην ομάδα εργασία βοήθησα του συναδέλφου για τη βοήθειά του. Ε, από το 2002 είμαι μέλος της Επιτροπής και μόνο βοήθεια είχα από τη γραμματεία, μόνο σεβασμό ένιωσα από τους συναδέλφους δεν είχα πρόβλημα ποτέ κανέναν. Με κανέναν. Από το 2002 που θητεύω στην Επιτροπή. Είχα ε, πολύ καλή συνεργασία. Και βλέπω μερικά μέλη της ομάδας μπροστά εδώ. Μπορεί να μην συμφωνούσαμε πάντα, αλλά με τη συζήτηση, με το διάλογο, με τη συνεννόηση, καταλήγαμε πάντα στη συμβαστική λύση. Μόνο συνεργασία και βοήθεια ε, γνώρισα σε όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στην Επιτροπή και σας ευχαριστώ όλους θερμά γι' αυτό. very kind words, so, uh, and thank you very much for uh, Πολύ όμορφα τα λόγια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική γνωμοδότηση που συντάξατε. Βλέπω ότι έχετε υποβάλει και κάποιες τροπολογίες για ορισμένα τμήματα τη γνωμοδότηση. Υπάρχει κάποιο που έχει αντίρρηση επί των τροπολογιών που έχει καταθέσει ο ίδιος ο εισηγητή. Όχι. Ωραία. Οπότε περνάμε στην ψηφοφορία ε, επί της ε, γνωμοδότηση αυτή. Παρακαλώ ψηφίστε. Okay, so now we can close the votes. Πέρα στις ψηφοφορίες. 171 ψήφοι υπέρ, μία αποχή. Συγχαρητήρια, κύριε Σίδα. Uh, Και με αυτό ολοκληρώσαμε το έργο μας για τις γνωμοδοτήσεις, αλλά πρέπει να εγκρίνουμε κάποιες αλλαγές που έγιναν κυρίως λόγω του ότι η Γκαμπριέλε Μπίσοφ, η συνάδελφός μας, έχει πλέον άλλα καθήκοντα ε, για τα οποία της ε, ευχόμαστε βεβαίως κάθε επιτυχία όπως επιτυχής ήταν και η δραστηριότητα της στην ΕΟΚΕ. Ο κύριος Ρούπκε λοιπόν αντικαθιστά την κυρία Μπίσοφ στο Προεδρείο της ΕΟΚΕ. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Η Ντόρτε Άντερσεν αντικαθιστά τον κύριο Βάντεγκαμπ στο Προεδρείο και πάλι, τον κύριο Βάντεγκαμπ που παρετήθηκε, δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσει. Ο κύριος Ρούπκε αντικαθιστά την κυρία Μπίσοβ ως μέλος της ομάδας σύνδεσης για την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ο κύριος Ρούπκε επίσης αντικαθιστά την κυρία Μπίσοφ στην, στην ε, στρογγυλή τράπεζα Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας και τέλος η κυρία Ογκορούρ θα αντικαταστήσει την κυρία Μπίσοφ στην ε, ομάδα εργασίας για τον εσωτερικό κανονισμό. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, οπότε εγκρίνεται και αυτή η αλλαγή. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη ζωηρή σας συμμετοχή στην ε, Σύνοδο Λομέλειας. Ολοκληρώνουμε το έργο, το έργο μας σήμερα. Η επόμενη ολομέλεια θα γίνει 15 και 16 Μαΐου στο κτίριο Σαρλεμάνι. Θέλω να σας ευχηθώ μια καλή μέρα και να ευχαριστήσω τη γραμματεία και τους διερμηνείς. Καλή σας μέρα. Γεια σας.